So, Καλώς ήρθατε όλοι στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πάνω. I will be chairing. Προεδρεύω. Δεμάς είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας για τη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και ξέπλυμα χρήματος και αντικαθιστώ τον κύριο Βέρνα Λάγκεν, τον πρόεδρό μας. Ο τίτλος λοιπόν της σημερινής συνεδριάσεως είναι ξέπλυμα χρήματος και φόρο αποφυγή. Ποιο είναι ο αντίκτυπο για τα κράτη-μέλη, πώ αποτελεσματικά τα κράτη-μέλη καταπολεμούν το φαινόμενο. Μόλι τώρα λάβαμε κάποιε μελέτε. Δεν μπορέσαμε να τι διαβάσουμε. impact presume, at least as a working Λοιπόν, μπορούμε να το επεξεργαστούμε το θέμα λοιπόν. Στην ημερήσια διάταξη Έχουμε πρώτα την έγκριση αυτής. Απεστάλλητε κάτι 8 Απριλίου 2017 στα μέλη. Έχετε σχόλια για την ημερήσια διάταξη. Ουχή. Οπότε πάμε στο δεύτερο σημείο που είναι ανακοινώσει του Προέδρου. Θα καλωσορίσω τα μέλη και το ακροατήριο. Έχουμε και αναμετάδοση στο διαδίκτυο, νομίζω. Σκοπός συνεδριάσεως είναι να παρουσιάσουμε ένα, τύπο, ένα κομμάτι της πανεπιστημιακής έρευνας που ανετέθη την Επιτροπή μας. Είναι πολύ καλό αυτό, διότι κάποια από τα μέλη μας ε, είχαν πολύ μακρά συνεδρίαση ψηφοφορία σήμερα, δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς, αλλά όταν διαρκεί πολύ ψηφοφορία, εμένα μειώνονται οι εγκεφαλικές μου δραστηριότητε. Και τώρα είναι ευκαιρία να τις αυξήσουμε τις δραστηριότητε. Είχαμε παρόμοια συνεδρίαση όπως η σημερινή στις 2 Μαΐου θα έχουμε κάποια πονήματα ήδη έχουν παρουσιαστεί σε πρώτερες ευκαιρίες και θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα της εργασίας αυτές. Αυτές οι μελέτες αντιπροσωπεύουν ένα βασικό κομμάτι ε, τη συλλογή στοιχείων ε, που συνέλεξε η Επιτροπή Εξεταστική. Σημερινή συνεδρίαση έχουμε τρεις μελέτες που θα παρουσιαστούν. Σωστά, μου λέει και η γραμματεία, υποδιαιρείται σε δύο πάνελ η συνεδρίαση. Πρώτο πάνελ. Ποιο είναι αντίκτυπο ε, τη φοροδιαφυγή, νομοποίηση παρανόμων εσόδων, εσόδων παράνομων δραστηριότητε, στα οικονομικά των κρατών μελών. Δεύτερο πάνελ, δύο μελέτε που εστιάζονται στο ρόλο που παίζουν τα κράτη-μέλη, ειδική κυβερνήση των κρατών μελών στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγή και της νομοποίηση παρανόμων εσόδων. Πριν ξεκινήσω επεξήγηση τη διαδικασία θα ακολουθήσουμε και πριν σα παρουσιάσω του ομιλητέ για την πρώτη μελέτη, θα σα δείξουμε και μια ταινιούλα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 These studies will hopefully help to design sound evidence-based policies and improve the welfare of EU citizens. Very well. Uh, we can see the progress. Καλώς βλέπουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Επιτροπή μας, διότι στην αρχή των Επιτροπών είχαμε τεχνικά προβλήματα και τώρα όλα πήγανε ρολόι με το βίντεο. Κάτι είναι και αυτό. Αντιμετωπίζουμε μεγάλη ανασφάλεια όσον αφορά τα στοιχεία για τον, τις απώλειες φορολογικών εισοδημάτων λόγω φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και του, της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων. Άρα αυτές οι μελέτες μου πολύ. Ως παρουσιάστηκαν τα πράγματα, στο δεύτερο πάνελ θα συζητήσουμε τις νομικές συνέπειες για τα κράτη-μέλη και Εκεί θα προβώσω κάποιο σύντομο σχόλιο. Στείλαμε ερωτηματολόγιο σε όλα τα μελη Να μας πούν ποια μέτρα πήραν. Αυτό αφορά τις μελέτες του δεύτερου πάνελ. Μέχρι τώρα δεν λάβαμε απαντήσεις από τη Μάλτα ούτε από την Ουγγαρία. Λυπηρό. Διότι έχει και την Προεδρία μάλιστα τώρα η Μάλτα του Συμβουλίου και θέλουμε να ενθαρρύνουμε να μας απαντήσουν δεν λάβαμε απαντήσει ούτε από τη Δανία ούτε από την Ισπανία, αλλά είπαν και οι δύο χώρε ότι συντομότατα θα απαντήσουν. Κάθε παρουσίαση μελέτη θα κρατήσει το πολύ 25 λεπτά. Άρα, οι τρει συνάδελφοι θα έχουν περίπου 7 λεπτά ο καθένας. Μετά τα δύο πάνελ θα γίνει ανταλλαγή απόψεων. Θα συμμετάσχουμε μέλη τη επιτροπή μα. Θα υποβληθούν ερωτήσει κανά πεντά λεπτά και απάντηση ένα λεπτό, ο υπόλοιπο χρόνο θα αφιερώνεται στην απάντηση. Αν υπάρχει χρόνο, θα μπορεί να, να ζητήσει να, κάποια διευκρίνηση ένα μέλο. Κάθε φορά πρέπει να. Όταν πατάει το, για να ανάψει το μικρόφωνο, ο μιλητή στρέφεται η κάμερα πάνω του, οπότε είναι χρήσιμο το ξέρετε αυτό. Πάμε στην πρώτη μελέτη. Αντίκτυπο των όσων αποκαλύφθηκαν από τα Panama Papers για τα οικονομικά των κρατών μελών. Έχουμε τον Mike Beek, εξεβονίμων. Τον David Buck στο μέσο και τον Jack Milan από το Κέντρο Υπηρεσιών Στρατηγικής εξολογήσεω. Και είναι υπεύθυνο ο Ζαν είναι από το τμήμα αναλύσεων. Πρώτα θα αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των φορολογικών παραδείσεων και των υπερακτίων περιοχών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη από πλευρά οικονομική, δημοσιονομική, χρηματοπιστωτική. Υπενθυμίζει τη βασική νομοθεσία που ισχύει στην Ευρώπη για αυτά και στον υπόλοιπο κόσμο, για να περιοριστεί ο αντίκτυπο των φορολογικών παραδείσεων και των υπερακτίων περιοχών και προτείνει μια σειρά κανόνων, ούτω ώστε να ενισχυθεί η τρέχουσα νομοθεσία, ούτω ώστε να καταπολεμηθεί καλύτερα η αρνητική συνέπεια των φορολογικών παραδείσεων. Η μελέτη επεστάλλει στα μέρη τη 18 Απριλίου του 2017 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΑ. Βλέπω τώρα, κοιτώ προ του ερευνητές μας. Α, εσύ θα πάρετε τον πρώτο, πρώτο λόγο. Α, εσείς. Έχετε το λόγο, λοιπόν. Πατήστε το κουμπί, ε. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε για να παρουσιάσουμε τη μελέτη για τον αντίκτυπο που έχουν τα διάφορα σχέδια και σχήματα που απεκάλυψαν τα Panama Papers για την οικονομία και τα χρηματοστατικά για τα κρατη μέλη. Τρεις από εμά θα με την παρουσίαση. Εγώ θα δώσω τον ακτήριο λάκτισμα και ο Ντέιβιτ θα συνεχίσει τον αγώνα και μετά ο Μάικ ε, θα κλείσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω μέσω επισκοπήσεως των στόχων που καλύπτονται τη μελέτη. Πρώτος στόχος. Τα ποσά που δεν εισραίουν στον προπολογισμό των κρατών μελών λόγω των όσων αποκαλύπτονται από τα Panama Papers. Μετά, εξετάζουμε κάτι άλλο, τις οικονομικές συνέπειες αυτών, δηλαδή της μη ροής των πόρων που δεν μπορούν να δαπανηθούν για προγράμματα και δραστηριότητε. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά, να δημιουργήσουν θέσει απασχόληση και πλούτου. Τρίτο τομέα. Αντίκτυπο αυτών που απεκαλύφθησαν από τα Panama Papers όσον αφορά το, χρη... το έγκλημα στο χρηματοδοτικό τομέα και πώς επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών συστημάτων. Να ευθύ εξ αρχής το εξή. Στην έρευνά μας εστιαστήκαμε στο βαθμό του δυνατού στα διάφορα κόλπα που χρησιμοποιούν άτομα για φοροαποφυγή. Δεν εξετάζουμε τις επιχειρήσεις. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο τομέων δεν είναι πολύ ξεκάθαρη βέβαια, διότι τα άτομα χρησιμοποιούν εικονικέ επιχειρήσεις κλπ. για να αποφύγουν το φόρο. Εμείς εστιαστήκαμε στο πώ τα κόλπα που αποκαλύπτουν τα Panama Papers βοήθησαν οι να αποφύγουν τους ε, φόρους και ποιε είναι οι συνέπειε όλου αυτού. Τρίτο στόχος που βλέπετε και στη διαφάνεια στο κάτω μέρος. ποια μέτρα υφίστανται και ποια μέτρα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν βάσει των υφισταμένων και ποιος μηχανισμός θα μπορούσε να καταπολεμήσει αυτές τις ε, πρακτικές. Τώρα στρέφομαι προς τη μεθοδολογία. Ουσιαστικά πρέπει να πρόκειται. Ακολουθήσαμε δύο προσεγγίσεις. Προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε τα οικονομικά αποτελέσματα, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των διαφόρων τεχνασμάτων που χρησιμοποιούνται. Πρώτα ακολουθήσαμε εμπειρική προσέγγιση. Κάναμε συνεντεύξεις και τέτοιου είδους παρεμφερεί έρευνε. σε έξι κράτη-μέλη που παρατίθενται Κύπρο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και Έγιναν εκτενείς συζητήσει με τις εθνικές αρχές, είχαμε και γραπτές συνεισφορές από διάφορες τέτοιες αρχές, πανεπιστημιακοί συνέβαλαν, εμπειρογνώμονες, δημοσιογράφοι, μας βοήθησαν να αποκαλύψουμε όλα αυτά τα τεχνάσματα. Δεύτερη προσέγγιση. Προσπαθήσαμε να παραγάγουμε εκτιμήσεις όσον αφορά τις δημοσιονομικές και οικονομικές συνέπειες χρησιμοποιώντας οικονομετρικές μεθόδους. Αυτό το έκανε ένας εμπειρογνώμων που ανήκει στην ομάδα μας. Χρησιμοποίησε την βάση δεδομένων όπους. Προσπάθησε να δει ποιες εταιρείε και άτομα εμπλέκονται στις καταθέσεις σε φορολογικούς παραδείσους και μετά έγινε μια σύγκριση με επιχειρήσεις που δεν εμπλέκονται σε αυτά τα τεχνάσματα και συνήγαγαν κάποια συμπεράσματα. Στη συζητήση θα μπούμε σε κάποιες λεπτομέρειες της μεθόδου που ακολουθήσαμε. Συναθρήσαμε τα πορίσματα στην έκθεσή μας και χαίρομαι να πω ότι οι δύο μέθοδοι που χρησιμοποίησαμε οδήγησαν σε εκτιμήσεις που ε, ταιριάζουν η μία με την άλλη. Μέσω δύο διαφορετικών μεθόδων καταλήξαμε σε παρόμοια αποτελέσματα. Τελειώνοντας τώρα, η έκθεση που έχετε υποδιαιρείται σε πέντε τμήματα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες διότι πιθανότατα είχατε δυνατότητα να ρίξετε ματιά. Τα πρώτα τρία τμήματα αυτής εξετάζουν το όλο πλαίσιο στο οποίο γίνονται οι δραστηριότητες. Φορο... Ε, υπεράκτια, οικονομικά κέντρα, φορολογική παράδειση κλπ. Και πήραμε και τι υφιστάμενε μελέτες να δούμε ποια είναι η κλίμακα των δραστηριοτήτων, ποιες πρακτικέ ακολουθούνται, να τα λάβουμε αυτά υπόψη. Στο τέταρτο τμήμα βάζουμε τα αποτελέσματα των δικών μα ερευνών και προσπαθούμε να δούμε οικονομικές και δημοσιομικές και άλλες συνέπειες των όλων τεχνασμάτων που αποκαλύφθηκαν από τα Panama Papers και συγκεντρωνόμαστε επί των πορισμάτων αυτού του σημείου στην παρουσίασή μας. Τελικό τμήμα, όπως προενέφερα, αναθεωρεί τις πρωτοβουλίες που υφίστανται και αναπτύσσει και κάποιες συστάσεις περί ενισχύσεως αυτών και περαιτέρω εξελίξεων των. Θα δώσω τη σκητάλη στον συνάδελφο τον Ντέιβιτ. Θα αναφερθεί στις επόμενες δύο διαφάνειες περί του πώς εξετάσαμε το θέμα των ποσών που στερούνται οι προπολογισμοί των κρατών λόγω, λόγω της χρήσης αυτών των τεχνασμάτων. Καλησπέρα και από μένα. Για να δούμε ποιες είναι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις πρέπει να καθορίσουμε πώς ακριβώς χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά στις χώρες μέλη είδαμε ότι στην περίπτωση των Panama Papers επρόκειτο κυρίως για άτομα, για ιδιώτε. Βλέπετε εδώ στον ε, πίνακα το ποσό το οποίο θα πρέπει να πληρωθεί, αλλά δεν πληρώνεται στις ε, χώρες μέλη ή πληρώνεται αργότερα. Όπως βλέπετε από την ε, διαφάνεια αυτά που φάνηκαν από τα συστήματα στο Panama Papers υπάρχει μη συμμόρφωση είτε μέσω φόρο αποφυγής είτε μέσω φόρο και επικεντρωνόμαστε, όπως είπαμε, στους ιδιώτες. Δεν μιλάμε εδώ για πολυεθνικές επιχειρήσεις ή για μεγάλες εταιρείες. Από τα στοιχεία που έχουμε λοιπόν σε εθνικό επίπεδο είναι αυτά τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει. Διαπιστώσαμε ότι τέτοια συστήματα μειώνουν τις ε, χρηματικές πηγές που μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους οι χώρες ε, μέλη. 88 εκατομμύρια λιγότερο το 2015 για παράδειγμα με μείωση 90 δισεκατομμύρια σε μερικές μόνο χώρες. Αν αυτό το δούμε συνολικά, αυτό σημαίνει ότι και από την περίπτωση των εγγράφων του Παρμά και από άλλες περίπτωση υπάρχει απώλεια πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Και αυτό αντιστοιχεί με τις εκτιμήσεις που έχουν κάνει διάφορες χώρες μέλη. 10 με 15% της όλους σκιώδους οικονομίας. Έτσι όπως έχει εκτιμηθεί από το 2011 που ήταν στο 1-3. Αυτό το 1-3 περιλαμβάνει τους ε, ε, παραδείσους οικονομικούς που έχουν χρησιμοποιήσει και ιδιώτες και εταιρείε. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω στον άδερφο το λόγο για να σας μιλήσει περισσότερο για τις επιπτώσεις τις οικονομικές. Ευχαριστώ, Ντέβιτ. Όπως ακούσαμε, οι δημοσιονομικές ε, επιπτώσεις για χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί αλλού, στην εκπαίδευση, στην υγεία, αλλά και σε άλλου τομεί, στη δημιουργία θέσεων απασχόληση, για παράδειγμα, στήριξη επιχειρήσεων, ε, επενδύσει σε υποδομές, μεταφορές ή σε μέτρα υπέρ των περιφερειών. Όσον αφορά την απασχόληση πιο συγκεκριμένα, είναι δύσκολο βέβαια να εκτιμήσει κανείς τις επιπτώσεις από τις εκτιμούμενες απώλειες από τα φορολογικά έσοδα στις χώρες μέλη, μια συντηρητική εκτίμηση θα ήταν γύρω στο 1,5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης που θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί από τα χρήματα αυτά τα οποία τελικά χάθηκαν. Βέβαια, δεν λέω ότι τα χρήματα αυτά έχουν απόλυτη αντιστοιχεία με τις θέσεις απασχόλησης αλλά αν μη τι άλλο, αν είχαν πάει τα χρήματα αυτά σε πολιτικές ε, υπέρ της εργασίας, σίγουρα θα είχαν τεράστιες επιπτώσεις και άρα η απώλεια αυτών των χρημάτων επηρεάζει πάρα πολύ τα διασυνομικά μιας χώρας. Είπαμε, θα μπορούσαν να είχαν βοηθηθεί άνεργοι, κυρίως μετά την κρίση που αυξήθηκε η ανεργία και αντιστοιχεί Όντω τι παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να είχαν γίνει στην εργασία. Τώρα γενικότερα, τι σημαίνει η παρουσία των ε, φορολογικών αυτών ε, παραδείσων στον δημόσιο τον ιδιωτικό τομέα. Ουσιαστικά τα χρήματα αυτά βγαίνουν από την πραγματική οικονομία και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία των κεφαλαίων. Στρεβλώνεται επίσης και ο ανταγωνισμός μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούν την αγορά. Από τα στοιχεία που έχουμε πάντως φαίνεται ότι υπάρχει πράγματι στρέβλωση από τους φορολογικούς παραδείσους. Πρώτα απ' όλα επειδή υπάρχει το απόρριτο, την πιστευτικότητα μέσα στην οποία λειτουργούν, οπότε υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες λείπουν από το κοινό, ενώ θα έπρεπε να τις είχε το κοινό, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αγορά. Επίσης, η έρευνά μας δείχνει ότι και οι επενδύσεις ε, πλήττονται γιατί υπάρχει ένας ασύμετρος κίνδυνος. Και το αποτέλεσμα είναι ότι χρειάζεται πιο ψηλή απόδοση των ε, επενδύσεων στην περίπτωση που έχουμε την απώλεια αυτή από τους φορολογικούς παραδείσους. Τώρα, αν οι πληροφορίε αυτές για τους φορολογικού παραδείσους γίνονται γνωστές, όπω έγινε σε αυτή την περίπτωση, υπολογίσαμε ότι η διαρροή ήταν 150 δις σε δολάρια σε κεφαλοποίηση για 1762 περιπτώσεις εταιριών που χρησιμοποιούσαν ε, δικά τους μέσα ειδικού σκοπού. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι έπεσε η τιμή για τις επιχειρήσεις εκείνες που είχαν ε, εξωχώριες δραστηριότητες και που λειτουργούσαν μέσα στο απόρριτο. Επηρεάστηκε αρνητικά η οικονομική παραγωγή επίσης στις χώρες εκείνες όπου είχαν συμφέροντα αυτές οι επιχειρήσεις. Όσον αφορά λοιπόν τις επιπτώσεις αυτές πάντα, βλέπουμε ότι η χρήση των συστημάτων αυτό που χρησιμοποιήθηκαν στα έγγραφα του Παναμά έχουν να κάνουν όχι μόνο με την φοροδιαφυγή, έχουν να κάνουν και με περιπτώσεις άλλης διαφθοράς, δωροδοκία, τρομοκρατία, ναρκωτικά, εμπόριο ανθρώπων, παράνομη μετανάστευση, έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Έτσι, οι αρχές άρχισαν έρευνες για φοροδιαφυγή παντού στον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει σχέση ανάμεσα στη χρήση τέτοιων εξωχώριων περιοχών και του οικονομικού εγκλήματος. Ακόμα περισσότερο όταν κοιτάμε τις διατάξεις συμμόρφωσης. Βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοια μέσα ειδικού σκοπού για την δωροδοκία και έτσι να μπορούν να κερδίζουν πολύ ε, μεγάλες συμβάσεις δωροδοκία, δηλαδή δωροδοκία αξιωματούχων επίσης. Άρα είναι μια παραβίαση που οδηγεί στην ε, διαφθορά με τη χρήση αυτών των μέσων ειδικού σκοπού. Και η ιστορία αυτή έχει επιπτώσεις εφόσον υπάρχουν κυρώσει, να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τέτοια μέσα επιχειρήσεις για δωροδοκία. Από τη Europol το 2010 ξέρουμε ότι 250.000 περιπτώσεις νομοποίησης παράνομου χρήματος εκδικάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε άλλη ακρόαση εδώ, η Europol είπε ότι 3.500 ε, αντιστοιχίες βρέθηκαν μεταξύ διαφόρων μορφών εγκλήματος. Πολλέ από αυτέ ήταν από χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που τις κατήγγειλαν για νομοποίηση παράνομου χρήματος. Τελικά πρόκειται για ένα ποσοστό όμω, το οποίο τουλάχιστον όσον αφορά τα έγγραφα του Παναμά δεν επηρεάζει τόσο πολύ τη γενική κατάσταση. Αναφέρονται πολλά ονόματα στους καταλόγους των εγγράφων του Παναμά. Το 2013 36.000 εγκληματικές οργανώσεις αναφέρονται. 388 ονόματα επίσης συνδέονται με δραστηριότητες ΦΠΑ. με απώλειες 100 δισεκατομμυρίων όσον αφορά την φοροδιαφυγή από το ΦΠΑ. Τώρα για το Ισλαμικό ε, την Ισλαμική τρομοκρατία, 13% ήταν οι περιπτώσεις που είχαμε με τέτοιε υπόνοιε. Γενικά μιλώντα τα ποσά αυτά, βέβαια τα νούμερα αυτά, πρέπει κανεί να τα ερμηνεύει με ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί οι αντιστοιχείς αυτέ τη ε, Europol δεν έχουν ακόμα επαρκώ ε, εξεταστεί και άρα δεν μπορούμε να βγάλουμε σίγουρα αποτελέσματα. Επίσης δεν είναι και πλήρη τα στοιχεία που έχει η Europol. Το τρίτο που αφορά τις, αφορά τις συστάσεις μας. Συστάσεις που έχουν γίνει βέβαια και παλιότερα εδώ στην Επιτροπή, αλλά τις επαναλαμβάνουμε. Πρέπει να επεταχυθούν οι έρευνες που γίνονται στις χώρες μέλη. Η πρώτη μας λοιπόν σύσταση βασική είναι να εγγυθούμε την προστασία των καταγγελόντων που εμπλέκονται σε περιπτώσεις τέτοιας φόρου αποφυγής. Πρέπει να υπάρχουν μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ανθρώπων αυτών. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της δικαιοσύνης που παίζει εδώ, είναι ότι έτσι θα έχουμε πληροφορίες διαθέσιμες και θα έχουμε και δεδομένα ποιότητας, πληροφορίες ποιότητας. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να προστατεύονται οι καταγγέλλοντες. Αλλιώς οι πληροφορίες θα κυκλοφορούν στα μυστικά και θα στρεβλώνονται. Το δεύτερο, δεύτερο... δεύτερο είναι ακριβώς η αποτροπή των ε, ατόμων ε, τα οποία θα κάνουν κάτι τέτοιο καθώς γνωρίζουν ότι υπάρχει δυνατότητα διαρροών και θα προστατεύονται οι καταγγέλντες. Ο ΣΑ μάλιστα το χρησιμοποιεί ως μέρος του σχεδίου του αλλά τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή διαφέρουν ε, όσον αφορά την προστασία των καταγγελόντων. Θεωρούμε όμως ότι αυτό το ζήτημα έχει σημαντικές επιπτώσεις και σε άλλους τομείς. Η δεύτερη σύσταση είναι να διατηρηθεί η πολιτική ουδετερότητα του ορισμού του φορολογικού παραδείσου. Το τονίζουμε αυτό για να προωθήσουμε την μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία. Γιατί βεβαίως ε, τα κριτήρια της συνεργασίας για να ορίζουμε τους καταλόγους αυτούς μπορεί βεβαίως, ε, μπορεί βεβαίως να ψήρουν κατηγορίες μεροληψίας. Προτείνουμε για λόγους ουδετερότητας να υπάρχει μια γκρίζα λίστα με ένα πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει και κράτη-μέλη της Ένωσης και τρίτες χώρες όπως υπάρχει ήδη ένα τέτοιο σχέδιο λίστας. Η τρίτη μας σύσταση είναι να προωθήσουμε την δημιουργια μητρωων μητρών πραγματικών ιδιοκτητών. Κάποια κράτη-μέλη κάνουν τέτοια μητρώα αυτή τη στιγμή και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημοσιεύσει έναν οδηγό βέλτιστων πρακτικών. οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και τα σχετικά με σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα μοιράζονται τις πληροφορίες για τους μετόχους και το ποσοστό τους. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι υπάρχουν διαφωνίες που αφορούν την ιδιωτικότητα και βέβαια η άλλη πτυχή είναι η χρήση κάποιων κοινών προδιαγραφών αναφοράς και βεβαίως το ότι θα σημαίνει αυτό για τις διοκτικές αρχές και συγκεκριμένα για την δίωξη και ανείχνευση περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Το τέταρτο, η τέταρτη σύσταση είναι μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να έχουμε αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα για το μέγεθος της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Γιατί έχουμε ακριβώς έλλειψη αξιόπιστων ε, δεδομένων και το έχει τονίσει αυτό η Κομισιόν το 2015 και έχει αρχίσει να συνεργάζεται με τη Eurostat και τα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί η συλλογή των δεδομένων. Η μελέτη αυτή τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες και βεβαίως το ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την εταιρική φοροαποφυγή και ε, φοροδιαφυγή και την ε, φοροδιαφυγή ατόμων όπου είναι πολύ ε, ελλειπή τα δεδομένα. Βεβαίω θα μπορούσε να λάβει αυτό διάφορες ε, μορφές. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο για, στον συνάδελφο για να συνεχίσει με τις ε, συστάσεις. Νομίζω ότι έχουμε λίγα λεπτά, οπότε δεν θα μπω σε λεπτομέρειε. Έχουμε τρεις άλλους, ε, τρία άλλα κριτήρια. να συνδεθούν περισσότεροι πληροφορίε κατά του ξεπλήματο χρήματο με την φορολογική διαφάνεια, να υπάρχει ακαιρεότητα και διαφάνεια χρητού χρηματοπιστωτικού τομέα και τέλο να αναλάβουμε πρωτοβουλίε για να ενθαρρύνουμε προδιαγραφέ ε, χρηστή διοίκηση, ε, χρηστή φορολογική διοίκηση. Να συνοψίσω πριν κάνουμε τη συζήτησή μα το εξή. Νομίζω ότι είναι δύσκολο για εμάς να ποσοτικοποιήσουμε τα μέτρα αυτά για τα οποία μιλούσαμε. Δηλαδή τα αποτελέσματα τέτοιων συστημάτων που αποκαλύφθηκαν από το Panama Papers στους περιβολισμούς των κρατών μελών και τις οικονομίες τους. Δύσκολο, γιατί οι πληροφορίες είναι κατακερματισμένες και δεν μας δίνουν μια πλήρη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σχετικά έχουμε μια αρκετά καλή πεποίθηση ότι έχουμε μια ένδειξη της κλίμακας ε, των συνεπειών αυτών των συστημάτων και είναι σαφές νομίζω από τους αριθμούς ότι μιλάμε για ουσιαστικό αντίκτυπο με μεγάλη κλίμακα θεωρούμε ότι θα χρειαστεί καιρός ε, για να βρούμε το τι συμβαίνει με αυτά τα συστήματα τύπου Panama Papers. Έχουμε απλά δει την κορυφή του παγόβουνου. Αλλά υπάρχουν μέτρα κατά την απόψή μας μπορούμε να λάβουμε τώρα για να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και προφανώς ευχαριστώ να απαντήσουμε τυχόν ερωτήσεις που έχετε. Thank Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Τηρήσατε ακριβώς το χρονοδιάγραμμα. insecurities when dealing with those. Υπάρχουν μεγάλες ανασφάλειες όσον αφορά τα στοιχεία. Στα έγγραφα του Παναμά είδαμε μόλις ένα κομμάτι των υπερχωρίων αυτών δραστηριοτήτων. Και δείχνουν ότι θα έχουν αντίκτυπο σε επενδύσεις, στην απασχόληση. Και ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον που είδατε στη βάση δεδομένων της Europol ε, Έχουμε και σημαντικές αποκαλύψεις γιατί τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την Ισλαμιστική τρομοκρατία. Πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό, εξετάζοντα αντιδράσεις των κρατών μελών, όπως το πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών. Καλά κάτω μας υπενθυμίστε κάποιες συστάσεις του Κοινοβουλίου, όπως η προστασία των καταγγελόντων είναι πολύ καλό να επαναλαμβάνουμε τις συστάσεις. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι γνωρίζω, ακόμα δεν έχει κινηθεί καταλήλως. Αρκετά αυτά που είπα. Ας πάρουν ε, οι συγητές πάνω και μετά τα υπόλοιπα μέλη. Η κυρία Κόφορτ των Σοσιαλιστών. Πέντε λεπτά. Πίτερ Τζέσεκ για την Άλντε. Ο Πίτερ, ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε τους ερευνητές και τους ακαδημαϊκούς Χρησιμότατα τα πορίσματα. Και χάρηκα για τελευταία σας σχόλια. Πράγματι έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για τα 19 δις για τα κράτη-μέλη, κάποια κράτη-μέλη, 100 εκατομμύρια ευρώ σε όλα τα κράτη-μέλη. Χαμένα έσοδα. Και θα μπορούσαν να, να είχαν δημιουργηθεί 1,5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Και αυτό είναι μόνο σε ατομικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο, ποιες είναι συνέπειες του προβλήματος. Φορολογική παράδοση, ε, υπεράκτια κέντρα κλπ. Στους ορισμούς θα να κινηθώ. Στο σημείο 2-3 είπατε πρέπει να υπάρχει πολιτική ουδετερότητα όσον αφορά τον ορισμό των φορολογικών παραδείσων. Η φορολογική παράδειση χρησιμοποιούνται από τους μεσάζοντες μέσα στο θολό αυτό τοπίο επιχειρήσεων και φορέων. Διευκρινήσεις παρακαλώ. Ποιους βασικούς δείκτες διαπιστώσατε στην ερευνά σας ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να καθορίσουμε φορολογικούς παραδείσους. Μπορείτε να επεκταθείτε από αυτού, ξέρω ότι είναι δύσκολο, σημαντικό. Δεύτερον, κάτι σχετικό. Ποια είναι η άποψή σας Ποιο είναι το βέλτιστο κριτήριο για τους φορολογικούς παραδείσους. Μετά. Κάντε κάποιες αξιολογήσεις. Σε οχτω κράτη-μέλη. Ανακαλύψατε δυναμίες σε μία από τις οκτώ χώρες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν οι δυναμίες της εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο των φορολογικών παραδείσων και των υπερχωρίων περιοχών. Είναι οχτώ χώρες διαφορετικές βέβαια. Ισχυρά και ασθενή σημεία των χωρών. Μπορείτε να μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα που μας σχεδιάσατε. Um, Πρώτη ερώτηση. Ορισμός φορολογικού παραδείσου. Έχουμε φορολογικό παράδεισο και υπερχώριο χρηματοστικό κέντρο. Φορολογικός παράδεισος. Έχουμε ορισμό των 98 του ΟΑΣΕ. Του ΟΣΑ, συγγνώμη. Που περιέχει κάποια χαρακτηριστικά για το φορολογικό παράδεισο. Πρώτον, αν χρησιμοποιούν ονομαστικού φόρου ή μη φόρου, όσον αφορά το εισόδημα, την κληρονομιά ή εταιρικό φόρο στου μη μόνιμου κατοίκου είναι όμως που εμποδίζουν την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών με κυβερνήσει και για τους φορολογωμένους. Τρίτον, αν λείπει η διαφάνεια στον φορολόγηση. Αν είναι πιο δύσκολο δηλαδή οι χώρε καταγωγή να λάβουν αμυντικά μέτρα ή να διώξουν, να ασκήσουν δίωξη για τη χρήση αυτών των μηχανισμών. Εν συγκρίση με τα υπερχώρια χρηματοδοτικά κέντρα, ποια είναι η διαφορά. Έχουμε του δουνουτού ορισμό αυτών των υπερχωριών χρηματοδοτικών κέντρων έχουν αξία χρηματοστικών υπηρεσιών δυσανάλογη προς την αξία της εγχώριου οικονομίας. στο κριτήριο, το δεύτερο που τονίσατε. Οι συνάδελφοι θα επεκταθούν από αυτό. Τι λέμε, ότι είναι πιο εύκολο να προσμετρήσουμε την περίπτωση υπερχωρίου αυτού χρηματοπιστωτικού κέντρου, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει δυσανάλογη κίνηση σχέση με την εγχώρια οικονομία, παρά να ορίσουμε τον φορολογικό παράδεισο. Δύσκολο αυτό. Να δούμε πόσο χαμηλός είναι ο φόρος. Σε πρώτερες έρευνες δεν έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Διότι υπάρχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα στον αφορά την των φόρων. Και πώ καθορίζουμε το όριο κάτω από το οποίο ε, μια περιοχή θεωρείται φορολογικό παράδεισος. Για το δεύτερο τώρα ερώτημα βαθμό στον οποίο το δείγμα των 7 χωρών, λέει ο μιλητή, επηρεάζει τα πορίσματα της μελέτης και τα σχηρά σημεία και αδύνατα σημεία των χωρών. Το δείγμα ήταν καλό. Εγκάρσια διατομή, αν θέλετε, μια διατομή των κατών μελών. Και δείχνει τα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28. Γι' αυτό επιλέξαμε και το δείγμα αυτό. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Θεωρούμε ότι είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Όμως, είχαμε διαφορετικά ποσά πληροφοριών και δεδομένων από τις χώρες. Κάποιες χώρες έδωσαν αρκετά ποιοτικά στοιχεία και ποσότητα στοιχείων, άλλες όχι. Οι εκτιμήσεις όσον αφορά το δημοσιονομικό αντίκτυπο, παρόλο που βασίστηκε στην έρευνα στις 7 χώρες του δείγματος, βασιστήκαμε περισσότερο σε κάποιε αυτέ τι χώρε, τις μεγαλύτερες τη ομάδα. περισσότερο σε αυτέ από τι άλλε. Αυτό βέβαια έχει συνέπειε Όταν προσπαθούμε να κάνουμε προβολή των πορισμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 28. Πράγματι είχαμε αδυναμίες εξ αυτού όσον αφορά το δείγμα λόγω ελλείψεως στοιχείων. Δεν ξέρω αν θα προσθέσουν οι συνάδελφοι κάτι όσον αφορά ισχυρά σημεία και δυναμίες των χωρών. Αυτά είναι τα βασικά που ήθελα να τονίσω εγώ από τη δική μου πλευρά. δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Είδαμε τα 8 κράτη-μέλη του δείγματος. Πολλοί όροι επηρεάζουν την κατάσταση. Πολλά ισχυρά και αδύναμα σημεία που μπορεί να επηρεάσουν τι εκτιμήσεις. Διαφέρουν οι καταστάσεις σε κάθε χώρα. Παράδειγμα. Οι δημοσιογράφοι στην Ισπανία υπέβαλαν κάποιες αναφορές και είχε δώσει αμνηστία ε, χρηματοδοτιστική, οικονομική, φορολογική σε κάποιους ανθρώπους. Οπότε ο κόσμος έφερε χρήματα πίσω λόγω αμνηστίας. Είχε εντοπίσει τα ποσά αυτά η κυβέρνηση, αλλά διαπιστώθηκαν ότι πράγματι είχαν γίνει αυτές οι κινήσεις μέσω των εγγράφων του Παναμά. Ήταν ορατές οι μετακινήσεις. Άρα είδαμε εδώ ότι αυτό επηρέασε τις εκτιμήσεις. Να ένα παράδειγμα. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα περνάμε στο δεύτερο συνεισηγητή, αλλά ο Πίτερ θα πάρει το λόγο. Όχι. Ο κύριος Λουί Μισελ. Από την Άλντε που εκπροσωπεί την Επιτροπή ολόκληρη ουσιαστικά. Ναι, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να δούμε πότε θα έχουμε τα γαλλικά, Πρόεδρε. Γιατί, εντάξει, είμαι καθηγητής αγγλικών, αλλά εγώ θα ήθελα τη μελέτη να τη διαβάσω στα γαλλικά. Είναι θέμα αρχής και όλο και πιο συχνά αναγκαζόμαστε και δουλεύουμε εδώ στα αγγλικά. Ενώ η χώρα η οποία κυρίω μιλάει αυτή τη γλώσσα σε λίγο δεν θα είναι καν μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα έπρεπε να το δούμε αυτό και να φροντίσουμε για τα γαλλικά. Τέλο πάντων, τεχνικό ζήτημα. Λοιπόν, τώρα έχω κύριε Μαλά μια συγκεκριμένη ερώτηση να σα θέσω. Πρώτα απ' όλα, σημειώνω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής που χρησιμεύουν για παρετέρω προβληματισμό, αλλά για να είναι πραγματικά χρήσιμα και αξιόπιστα θα πρέπει οι βάσεις δεδομένων πάνω στις οποίες δουλέψατε να είναι αδιαφυσβήτητες. Οπότε ρωτάω, ξέρουμε ότι σε αυτό το πακέτο των Panama Papers ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια μοντάζ, μπορούμε να τα καθορίσουμε άνισα, ή μάλλον παράνομα που και άλλα που δεν είναι παράνομα. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ηθικά, αλλά δεν είναι και παράνομα. Οπότε ρωτάει, βάσει δεδομένων που χρησιμοποίησατε εσείς για τη μελέτη σας, είναι όλα ε, δεδομένα που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες ή εσείς ασχοληθήκατε συνολικά με όλες τις συναλλαγές χωρίς να μπορέσετε να κάνετε διάκριση ανάμεσα σε αυτά που ήταν παράνομα και αυτά που ήταν νόμιμα. Και η ερώτησή μου δεν είναι, πώς θα το πω, δεν την κάνω εκ του πονηρού καθόλου. Γιατί στη δικαιοσύνη αυτό θα παίξει ρόλο γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει ό,τι συστάσεις κάνετε να έχουν σαν βάση το δίκαιο. Για μένα λοιπόν είναι σημαντικό. Μα λόγια, εσείς εκτιμήσατε εμπειρικά από αυτά τα οποία επιλέξατε και βάσει αυτών καταλήξατε στα συμπεράσματά σας. Δεύτερον, φορολογική εναρμόνιση στην Ευρώπη. Δηλαδή να έχουμε τους ίδιους υπολογισμούς για τη φορολογία επιχειρήσεων παντού στην Ευρώπη. Είναι εφικτό. Όταν ξέρουμε τις συμφωνίες που γίνονται ανάμεσα στις κυβερνήσεις και τις πολυεθνικές έχουν αυξηθεί μετά το LuxLeaks. Και οι ρυθμίσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι πολλές και για να υπάρξει συμφωνία στο φορολογικό πρέπει να υπάρχει ομοφωνία στην Ευρώπη. Πώς θα γίνει λοιπόν. Ο έλεγχος θα ήταν καλός αν γίνεται στοχευμένα η... και για να υπάρξει πίεση σε όλες τις χώρες μέλη θα πρέπει να είναι γνωστή η φορολογική παράδειση. Εγώ έχω κάνει την ίδια ερώτηση σε όλους όσοι πέρασαν από εδώ και δεν πήρα απάντηση δεν τα βάζω μαζί τους, αλλά να, η ερώτηση είναι εξή. Τι διαφορά βλέπετε εσείς ανάμεσα στην έννοια ή τον ορισμό της φόρο αποφυγής, φόρο διαφυγής και της απόκρυψης. Υπάρχουν αποχρώσεις και πάνω στις αποχρώσεις αυτές παίζει κανείς και βασίζεται. Τώρα η εκτίμηση που γίνεται, και εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι και εύκολο, ρωτάω λοιπόν, εκτίμηση του διαφυγόντος κέρδους του φορολογικού υπάρχει για ολόκληρη την Ευρώπη Καταλαβαίνω ότι εσείς βασιστήκατε σε 8 χώρε, ναι, αλλά εκτό πέρα από αυτή τη μελέτη, υπάρχουν κάποιοι, ξέρω εγώ, στατιστικοί Ινστιτούτα έχουν δεδομένα για το σύνολο τη Ευρώπη. Και αυτή είναι μια ερώτηση που πιστεύω ότι είναι σημαντικό να απαντηθεί. Τέλος, έχω κάποιες αμφιβολίες για την απώλεια απασχόληση. Εσείς μιλάτε, λέτε 1,5 με 3,5 εκατομμύρια απώλεια θέσεων απασχόλησης όταν εσείς ε, τιμολογείτε 50.000 ευρώ μια θέση απασχόλησης. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι αυτό το κόστος, τουλάχιστον στη δικιά μου τη χώρα δεν ε, πιστεύω ότι κοστίζει τόσο το διπλά. 50.000, ίσως το δημόσιο ναι, αν είναι να κερδίσουμε τα χρήματα αυτά για να τα επενδύσουμε στο δημόσιο και να προσλάβουμε δημόσιους υπαλλήλους, αυτό είναι κάτι άλλο, έτσι, αλλά αυτό είναι πολιτική επιλογή. Είναι σημαντικό για την αξιοπιστία. Εγώ θα βάζα παραπάνω. Είναι πιο τεχνικό πάντως αυτό το ζήτημα του πόσο κοστολογείται μια θέση απασχόλησης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Μισελ, τα γαλλικά είναι μια πολύ σημαντική γλώσσα και πάρα πολύ όμορφη. Και είναι απόλυτα θεμητό να μιλάμε γαλλικά εδώ περίληψη υπάρχει στα γαλλικά, αλλά ολόκληρη μελέτη υπάρχει μόνο στα αγγλικά. Λοιπόν, για να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Ο κύριος Μαλάν. Ευχαριστώ. Θα ζητήσω από τους συναδέλφους να απαντήσουν σε 6-7 ερωτήσεις και εγώ θα επικεντρωθώ στις δύο τελευταίες. Θα προσπαθήσω να απαντήσω την πρώτη και ο Μάικ την δεύτερη για το θέμα της νομικής ε, διάκρισης, ε, φοροδιαφυγής ε, και φοροαποφυγής. Κοιτάξτε, είδαμε ακριβώς ποιο ήταν το φορολογικό κενό λόγω Panama Leaks και από φορο αποφυγή την νόμιμη και από φοροδιαφυγή δηλαδή την παράνομη δραστηριότητα. Και αντιλαμβανόμαστε, παραδείγματο χάρη, ότι σε κάποιο κράτος μέλος ε, το εθνικό πλαίσιο θα αναφέρει ε, μία εκτίμηση ε, με τις νόμιμες χρήσεις και κάποιο άλλο με τις παράνομες. Η διάκριση μεταξύ των δύο Δυσκολεύει ομολογουμένως το να εκτιμήσουμε τον συνολικό αντίκτυπο των Panama Papers ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το θέμα της δημιουργίας θέσεων εργασίας έχετε απόλυτο δίκιο γι' αυτό ακριβώς έμφαση πρέπει να δοθεί στην αγορά εργασίας ε, και τις παρεμβάσεις ε, στην αγορά εργασίας. Έχουμε κάνει μια πολύ συντηρητική ε, προσέγγιση και μια αναλογία ένα προς ένα. τώρα από ό,τι βλέπω από τα δεδομένα, για να δω, Παραδείγματο χάρη, αν ε, δούμε την οικονομική ανάπτυξη μεταξύ 2005 και 2008, είχαμε μείωση κατά 20% των ανέργων και οι δαπάνες ε, για μέτρα αγοράς εργασία μειώθηκαν. Αλλά με την οικονομική κρίση βλέπουμε ότι ε, αυξάνει το αριθμό των ανέργων και βεβαίως οι δαπάνες των κρατών για μέτρα αγοράς εργασίας αυξήθηκαν. Αυτή η αλλαγή λοιπόν το 2010 ε, είναι μεγάλη. Δηλαδή συνέχισε να ανεβαίνει ο αριθμός των ανέργων. Το 2011 οι δαπάνες για μέτρα αγοράς εργασίας μειώθηκαν ενώ ο αριθμός των ανέργων σταθεροποιήθηκε. Οπότε τα φορολογικά έσοδα. Αυτό προσπαθούμε να πούμε θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα κράτη να ασκήσουν πολιτική αγοράς εργασίας. Θα στήριζαν π.χ. 140.000 Ευρωπαίους πολίτες που έχασαν τη δουλειά τους το 2010-2011. για να ε, έχουμε έτσι μια ιδέα του αντικτύπου. να συμπληρώσω κάποια πράγματα κόστος ανά θέση εργασίας. Βγάλαμε ένα μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως γνωρίζω ότι σε κάποια κράτη-μέλη είναι πολύ ψηλότερος ο αριθμός από αυτόν που υπολογίσαμε. Αλλά αυτό νομίζαμε ότι θα είναι ο λογικός αριθμός για τα 28 κράτη. Για το θέμα των 8 χωρών και το αν θα υπήρχαν ε, δεδομένα για τις 28. ασχοληθήκαμε μόνο με κάποιες χώρες που δεν υπήρχαν στο δείγμα μας. Και δεν ε, πήγαμε πέρα από το δημοσίως διαθέσιμα υλικά. Ε, ο πρόεδρος, έχουμε ξεπεράσει λίγο το χρόνο και θα πρέπει λίγο να βιαστείτε. Ζητώ συγγνώμη, εγώ φταίω γιατί δεν είχα το εργαλείο εδώ, το χρονόμετρο. Οπότε τώρα το έχω. Ο επόμενος ομιλητής είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο κύριος Φάντεν Καντελάρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα που έχετε σφυράκι θα είμαι γρήγορος. Να ευχαριστήσω τους ερευνητές για την μελέτη αυτή που πραγματικά μας δείχνει ξεκάθαρα τα αποτελέσματα που μπορούν να έχουν για τον προϋπολογισμό και την οικονομία των κρατών μελών αυτές οι έρευνες και βεβαίως ε, να αντιμετωπίσουμε και τα πιθανά αδικήματα. Βεβαίως νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα προωθήσουμε αυτά για να ασχοληθούν περισσότερο τα κράτη-μέλη. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Έχω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτο είναι το εξής. Στην μελέτη σας μιλάτε θετικά για το ότι το Common reporting ε, standard ε, θα υιοθετηθεί από τους περισσότερους φορολογικούς παραδείσους. Βλέπουμε όμως ότι το πρόβλημα δεν αφορά τις επίσημες δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν η φορολογική παράδοση, αλλά η έλλειψη πραγματικής ε, εφαρμογής. Και ο Παναμάς είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οπότε το ερώτημα είναι πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ισχυρό εμπορικό μπλοκ να φροντίσει αυτά τα reporting standards και οι άλλες διεθνείς υποχρεώσεις να εφαρμόζονται πραγματικά. Δεύτερη ερώτηση, αναφέρεστε σωστά στην υποκρισία των ΙΠΑ που έχουν βεβαίω μια μονομερή πρακτική την οποία ακολουθούν όσον αφορά την μετάδοση δεδομένων ενώ προστατεύουν τους δικούς τους κατοίκους απέναντι σε εφορίες άλλων χωρών. Οπότε έχουμε ένα μια χώρα η οποία απειλεί να γίνει μια φορολογική μαύρη τρύπα, θα λέγαμε. Τι θα κάνουμε, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ε, φάτκα για τις χώρες οι οποίες δεν θέλουν να έχουν διαφάνεια. Όταν παραδείγματος χάρη ε, τα άτομα αυτά ε, βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, σας ευχαριστώ. Τρία λεπτά έχουμε για την απάντηση. Um, e uh, τι μορφή πρέπει να έχουν τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούμε. Από ό,τι κατάλαβα ότι χρειαζόμαστε κάποια, κάποια task force χρηματοπιστωτικής δράσης η μονάδα συλλογή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μυστικών πληροφοριών του ΣΥΠΗΝ. πώς πρέπει να βελτιώσουμε ανταλλαγή πληροφοριών και όχι μόνο ανταλλαγή, αλλά και την ποιότητα των πληροφοριών μεταξύ μονάδων. Αυτό θα έχει θετικά τα αποτελέσματα στην εσωτερική αγορά και το εμπόριο. Στι προσπάθειε μα μιλήσαμε με εκπροσώπου εθνικών αρχών και διαπιστώσαμε ότι πολύ συχνά όταν υπάρχει συνεργασία, υπάρχει συνεργασία και μοίρασμα πληροφοριών, αλλά δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο τυποποιημένο. Δεν αμφισβητείται όμω η χρησιμότητα ανταλλαγή πληροφοριών όταν αυτήν τη χάνη λαμβάνει μέρο. Έξοχα, λέει ο πρόεδρος. Συνάδελφε Κονφεράτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους φιλοξενούμενους για την συνεισφορά τους στις εργασίες μας. Μα ανακουφίζει το γεγονός ότι και εκείνοι στις έρευνες που διεξήγαγαν ενετόπισαν μια τάξη μεγέθους, μια διάσταση των πόρων που αφαιρούνται από τα κράτη-μέλη μέσω της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Η αφορά την ποσότητα των συνεπιών, όσον αφορά την απασχόληση, αυτό μπορεί να συζητηθεί και να αξιολογηθεί διαφορετικά. Όμως αντιμετωπίζουμε πάρα πολλούς πόρους, οι οποίοι σε μια περίοδο κρίσης που διαρκεί χρόνια, όπως η ευρωπαϊκή κρίση, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να παράγουν θετικά αποτελέσματα για τα κράτη-μέλη. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί σύνταξης καταλόγου χωρών που παραβαίνουν τους κανόνες των φορολογικών παραδείσων. Θα έπρεπε να περιοριστούμε, ε, δεν θα έπρεπε να περιοριστούμε στις χώρες, συμφωνώ με την πρότασή σα. να συμπεριλάβουμε στον κατάλογο αυτών προφανώς και ευρωπαϊκές χώρες. Η βοήθειά σας σε αυτόν τον τομέα είναι σημαντική για μας. Σω έχετε συγκεκριμένη άποψη για το ποιες ευρωπαϊκές χώρες βάσει των όσων γνωρίζουμε θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτόν τον κατάλογο των φορολογικών παραδείσων. Σε συνάρτηση με αυτή την πρώτη ερώτηση, θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψή σας σχετικά με το θέμα των κυρώσεων. Διότι μιλάμε λίγο, πολύ λίγο για τις κυρώσεις. Αν υφίσταται, αν υπάρχει μια χώρα που έχει τα χαρακτηριστικά, αυτά που περιγράψατε, ενός φορολογικού παραδείσου, Πώς μπορεί να τιμωρηθεί, ποια μέσα κατά την απόψή σας είναι τα αποτελεσματικότερα για να τιμωρηθεί η χώρα. Διότι αν εντοπίσουμε τον αμαρτωλό, αλλά δεν τον τιμωρήσουμε, ίσως είναι καθαρά ε, νοηματική άσκηση η προσπάθειά μας και δεν έχει συνέπειες κοινωνικές ή οικονομικές. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Τι κυρώς θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε. Είναι σημαντικό αυτό να το διαπιστώσουμε, να το εξετάσουμε μάλλον. Και βέβαια ευχαριστώ και τον για την απάντησή σας. Δυόμιση λεπτά λέει ο Λοιπόν, το θέμα του καταλόγου αυτού της μαύρης λίστας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τι μορφή θα πρέπει να έχει αυτή η δημοσίευση. Ποικίλει η προσέγγιση δεν είναι κάτι μανιχαϊστικό λευκό και βαύρο. Χρειάζεται μια γκρίζα λίστα να εντοπίσουμε ποιε χώρε συνεργάζονται και ποιε προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το θέμα. Άρα ουσιαστικά στην πράξη είναι φορολογική παράδειση. Και ποιε χώρε αγνοούν από την άλλη το θέμα και δεν κάνουν τίποτα. Έχουμε τέτοιε χώρε που αγνοούν την task force, τη δικαιοδοσία τη task force και έχουν μπει στον κατάλογο. Οπότε είναι θέμα, α πούμε, αυρική. Για τα κράτη-μέλη όμω Ευρωπαϊκή Ενώσεω πρέπει να εξετάζουμε. Κάνουν προσπάθεια ή δεν κάνουν προσπάθεια. Το Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματο χάρη, αναφέρεται στα Panama Papers, σαν φορολογικό παράδεισο. παράδεισος. Η μικροοικονομική αξιολόγηση δείχνει ότι υπάρχει απώλεια στι εθνικέ αρχέ. Αλλά ηγούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο δημοσιεύοντα μητρό πραγματικών ε, ιδιοκτητών και δικαιούχων ιδιοκτητών. Άρα δύσκολο αυτό για τι οικονομικέ κυρώσει. Το μοντέλο που συστήνουμε είναι να δώσουμε κίνητα για συνεργασία. Και εκεί χρησιμεύει μια γκρίζα λίστα. Ο ΩΣΑ το έκανε αυτό. Το έκανε το 2009 και το 2000. Δημοσίευσε μαύρες λίστες φορολογικών παραδείσων και αφαιρούσε δικαιοδοσίες βάσει συμπεφωνημένων διεθνών προδιαγραφών. Εάν συναυτούν τέτοιες διεθνείς συμφωνίες, θα ήταν κάτι καλό και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι σε καλή θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σμαλούκα, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνηθίζεται εδώ μέσα να είμαστε ευγενικοί και διπλωμάτες, αλλά εγώ θα ήθελα να πω ότι απογοητεύτηκα πολύ από αυτά που μας είπατε σήμερα εδώ. Τίποτα από αυτά τα οποία μας παρουσιάσετε σήμερα δεν είναι κάτι το καινούριο. Δεν μάθαμε τίποτα. Τα νούμερα μας λέτε, τα έχουμε δει στις εφημερίδες ήδη, δεν μάθαμε τίποτα λοιπόν για το πώς καταλήξετε σε αυτό το νούμερο. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα για το πώς γίνονται οικονομετρικές εκτιμήσεις με βάση αυτά τα οποία μας είπατε το τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει με δισεκατομμύρια ευρώ περισσεύουν ε, οι κασίες αυτές. Έτσι, με συγχωρείτε και θυμίζουν έτσι, τεχνισμό. και ο πρόεδρος είπε πάρα πολύ ευγενικά και διπλωματικά ότι μας είπατε αυτά τα οποία ήδη ξέραμε και δεν τα είχαμε ξεχάσει. Αυτά τα ξέραμε. Δεν υπήρχε τίποτα το οποίο εμβάθυνε. Δεν υπήρχε κάποια μεθοδολογία. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει καν να μεταφραστεί αυτή η μελέτη. Ειλικρινά, ε, εγώ σας λέω τουλάχιστον δεν έμαθα τίποτα από αυτό και δεν βλέπω το λόγο να μεταφράσουμε τη μελέτη σας σε άλλες γλώσσες. Υποθέτω ότι είναι θέμα δικαιοσύνης Ο καθένας εδώ έχει το δικαίωμα να πει τη γνώμη του επί της μελέτης, οπότε είναι θέμα δικαιοσύνης να επιτρέψουμε σε όλους. Και εσείς βεβαίως, αν θέλετε να απαντήσετε, βεβαίως θα σας δώσω το λόγο. Συγγνώμη αν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας η έκθεση, αλλά εμείς σαν εντολή είχαμε να εξετάσουμε τις επιπτώσεις του συστήματος αυτού των εγγράφων του Παναμά, τις επιπτώσεις στην, ε, στα οικονομικά και στα δημοσιονομικά. Κάνουμε μία εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων, όπως μας ζητήθηκε. Εξετάσαμε ευρέως τι έρευνες υπάρχουν, τι πληροφορίες ήταν διαθέσιμες. Ομολογώ ότι δεν υπήρχαν πολλές, στις διάφορες χώρες που εξετάσαμε καταφέραμε να έχουμε πρόσβαση και σε έγγραφα τα οποία δεν ήταν δημόσια και καταλήξαμε έτσι στις εκτιμήσεις μας. Τώρα για το δεύτερο στόχο χρησιμοποίησαμε την απασχόληση ως δίκτυ για να εκτιμήσουμε τις γενικότερες επιπτώσεις. δεν μπορούσαμε βέβαια με τα μέσα που διαθέταμε να κάνουμε μια πλήρη έρευνα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να λάβουμε υπόψη μας όλες τις επιπτώσεις και όλους τους παράγοντες που έχουν να κάνουν με τα Panama Papers. Αλλά οι επιπτώσεις στην απασχόληση έτσι κι αλλιώ πιστεύουμε ότι είναι σημαντικές και από εκεί προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε κάποιε άλλε εκτιμήσει. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει άλλη εκτίμηση προηγουμένω από τις, για τις επιπτώσεις των ε, σκανδάλων που αποκαλύφθηκαν με τα Panama Papers. Βάσει αυτών που μας ε, ζητήθηκε, καταλήξαμε σε εκτιμήσεις για να καλύψουμε αυτό το κοινό. Είπαμε από την αρχή, αυτό το κοινό, είπαμε από την αρχή ότι πρόκειται για εκτιμήσεις, ότι βασιζόμαστε σε ότι ήδη υπάρχει, έτσι κι αλλιώς, και τα σκεφτήκαμε κατά πολύ να δούμε μήπως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και κάτι παραπάνω, αλλά σε αυτό καταλήξαμε. Δεν νομίζω ότι θα θέλατε εμείς να εφεύρουμε καινούργια πράγματα τα οποία δεν ήταν γνωστά και να βασιστούμε σε τέτοια. Ε, Όντω ο κ. Φαλουκά είναι πάρα πολύ ευγενή συνάδελφο και νομίζω ότι συμφωνεί ότι δεν φταίνε οι ερευνητέ που παρουσιάζουν ξανά και ξανά τι ίδιε συστάσει. Εμεί είμαστε αυτοί που πρέπει να τι εφαρμόσουμε τι συστάσει αυτέ. Λοιπόν, Άλντε, δεν βλέπω κανεί να έχει ζητήσει το λόγο. Ο κ. Μισελ μίλησε ήδη. Οπότε, αν δεν διαμαρτύρεται η Άλντε, θα πάω κατευθείαν στην ΚΟΕ. Μακάρτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Έχουμε κάποια άποψη για διάφορα σημεία της έκθεσης. Εντάξει, συμφωνώ ότι είναι σημαντική έκθεση, αλλά μία από τις αδυναμίες είναι ακριβώς ότι τώρα μαθαίνει ο κόσμος όπου οφείλεται η απώλεια χρημάτων εξαιτία της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής κτλ. Αλλά δεν φτάνει να λέμε ότι αυτό ζημιώνει τις εθνικές οικονομίες. Είναι ένα ευρύτερο επιχείρημα. Και κάποιοι από εμά μπορεί να τα ξέρουμε τα ποσά, τα νούμερα. Οι περισσότεροι όμως πολίτες δεν το ξέρουν, γιατί βέβαια δεν διαβάζουν την κάθε έκθεση η οποία αναφέρει τη μεγάλη ζημιά πολιτική, οικονομική και κοινωνική που απορρέει από τέτοιες πρακτικές. Έχω μερικές σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη μου έχει να κάνει με το τμήμα της έκθεσης που αναφέρεται σε θεμητούς και αθέμητους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούνται εικονικές εταιρείε. Και που είναι το όριο ανάμεσα στο νόμο και το παράνομο αναφέρονται περιγραφές με φοροποφυγή εταιριών και ιδιωτών. Μπορείτε να μας περιγράψετε ποιες μπορεί να είναι οι νόμιμες χρήσεις τέτοιων εικονικών εταιριών που δεν οδήγησαν σε φοροποφυγή. Και επί τόσον αφορά το οικονομικό έγκλημα και εκτίμηση που κάνατε για αυτή την έκθεση. Η ερώτηση δηλαδή είναι τι δεδομένα πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε για να εντοπίσουμε ακριβώς τον οικονομικό αντίκτυπο από τα Panama Papers. Και άλλες δύο ερωτησούλες και με σύντομες απαντήσεις μπορείτε να μου απαντήσετε. Είπατε πολλές φορές ότι η διαφορά έγκυται στην ποιότητα πληροφοριών που έχετε από τις διάφορες χώρες. Ποια χώρα δεν σας έδωσε τις πληροφορίες που θα χρειαζόσασταν και τέλος, αναφερθήκατε στον ορισμό των φορολογικών παραδείσων. Ποια χώρα μέλος, αν υπάρχει καμία τέτοια, θα τέριαζε με αυτόν τον ορισμό που εσείς μας δώσατε. Θα, ήθελα να ζητήσω από τον Ντέιβιν να αναφερθεί σε αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, η έκθεση αυτή ε, δεν είναι εξαντλητική όσον αφορά τις εταιρείε αυτές, αλλά με την έννοια της σύστασης μιας νομικής οντότητας offshore ε, καθορίζεται αυτό από το πώς μεταφέρονται τα κέρδη και μέσω ποιών διάβλων. Οπότε εξετάζουμε μια εταιρεία που έχει συσταθεί αλλού και χρησιμοποιείται μέσω χρηματοδότησης χρέους είτε μέσω μετακίνησης ε, των ε, εσόδων ε, το κόστος σε άλλη δικαιοδοσία. Δεν εστιάσαμε τόσο στην διάκριση νόμιμου, παράνομου για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο στον προπολογισμό όπως είπα πριν. Για το είδος των δεδομένων που απαιτείται για να καθορίσουμε τον αντίκτυπο Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η έκταση του ξεπλήματος χρήματος είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή γιατί υπάρχουν πολλά γκρίζα νούμερα και πολλές περιπτώσεις δεν ανοιχνεύονται οπότε εκείνη τη στιγμή εξαρτάται κανείς από δεδομένα των περιπτώσεων που έχουν ανοιχνευθεί και συλλέγονται με διαφορετικό τρόπο έμειναν για δεδομένα που συλλέγονται στην φάση των πληροφοριών και μετά υπάρχει και η φάση της έρευνας. Οπότε, ε, το νούμερο που ανέφερε η Eurostat π.χ. 250.000 ε, περιπτώσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύσκολα συνδέεται με τα Panama Papers γιατί βεβαίως είναι και μόλις πριν από ένα έτος και οι περιπτώσεις αυτές συνήθως χρειάζονται πολλά χρόνια. Οπότε ίσως τα επόμενα χρόνια όταν θα μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε τις περιπτώσεις με τα δεδομένα θα είναι πιο σαφές το ποιες είναι οι σχέσεις δηλαδή. Αυτά. Να αναφέρω και εγώ να απαντήσω σύντομα στην τρίτη ερώτηση ποιες χώρες δεν έδωσαν δεδομένα. Είχαμε κάποια δεδομένα από όλες τις χώρες βεβαίως διαφορετικού τύπου δεδομένα και δεν είχαμε συγκεκριμένες ε, εκτιμήσεις για το ε, ποιοι ήταν οι διαφυγόντες φόροι π.χ. η Γερμανία και η Πολωνία δεν μπόρεσαν να το ποσοτικοποιήσουν οπότε έχουμε καλές πληροφορίες στις περισσότερες ε, χώρες αλλά όχι πάντα ποσοτικοποιημένες σας ευχαριστώ ο Σβέν Γκίγκολντ από τους Πράσινους Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα. Κοιτάξτε, σε κάποια φάση είχα παρόμοια ερώτηση, όπως ο κ. Λόκε. Δεν κατάλαβα κάτι. Πώς υπολογίσατε και βάσει ποιων στοιχείων τα στοιχεία σας. Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένοι. Πώς τα υπολογίσατε. Ποια μέθοδο χρησιμοποίησατε. Ποια ήταν η οικονομετρική σας προσέγγιση. Πώς διαφέρει η μεθοδολογία δική σας από τις άλλες μελέτες που κυκλοφορούν. Αυτό είναι το πρώτο που έχω να θέσω. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω το παντώντας. Στην αρχή είπαμε κάτι. Ακολουθήσαμε δύο μεθόδους στη μελέτη. Η μία εμπειρική. Τι κάναμε, πήγαμε στα κράτη-μέλη, ζητήσαμε πληροφορίες για τις φορολογικές απώλειες. Δεύτερη μέθοδος, οικονομετρικό μοντέλο. Δεν εδραστήκαμε αποκλειστικά από τις μία μεθόδους. Συνδυάσαμε τις δύο. Συλλογή στοιχείων στον εμπειρικό κλάδο της προσπάθειας. Ζητήσαμε τις αρχές να μας πούν πόσο εκτιμούσαν τη φορολογική απώλεια όταν δεν παίρναμε κάποια εκτίμηση, όπως σε κάποιες χώρες. Είδαμε τι γινόταν στις χώρες που μπορούσαμε να πάρουμε στοιχεία και κάναμε μια προβολή, αν θέλετε, και μια προσωμείωση και στις χώρες που δεν μας δίνουν στοιχεία. για το οικονομετρικό μοντέλο. Βασιστήκαμε στη βάση δεδομένων Orbis. Το ανέλαβε κάποιος που δουλεύει πολύ για την Επιτροπή. Εξέτασε δύο δείγματα. Περιπτώσεις όπου άτομα μέτοχοι σε εταιρείε που αναφέρονται στα έγγραφα του Παναμά είχαν εμπλακεί και περιπτώσεις όπου οι μέτοχοι και εταιρείε δεν είχαν αναμειχθεί σε αυτά που αποκάλυψαν τα έγγραφα του Παναμά. Κάναμε σύγκριση των δύο δειγμάτων λοιπόν. Και από την σύγκριση προέκυψε το μοντέλο και εκτιμήσεις για τα κέρδη και τους φόρους και τι ποσό θα μπορούσε να εμπλέκεται στις μεθόδους φόρα που θα δώσουν περισσότερες πληροφορίες και για τα όσα κάναμε μέσω της εμπειρικής προσεγγίσεως, μέσω των συνεντεύξεων και της συλλογή στοιχείων από το δείγμα κρατών μελών και για το οικονομετρικό μοντέλο. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες πληροφορίες που δεν στην έκθεση. Βλέπαμε ότι δεν θα ενδιαφερόταν πολύ για αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες για το οικονομετρικό μοντέλο. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θα να προσθέσει. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Μάλλον ο κ. Ζήκο για τι συμπληρωματικέ πληροφορίε που θα μα στείλετε για το οικονομετρικό μοντέλο, για το πρώτο κομμάτι. Σωστά το εκλαμβάνω. Αθήσατε στοιχεία που πήρατε από εθνικέ αρχές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους περί φορολογικών απολειών που απέρα από διαφορετικές μεθοδολογίε, διαφορετικού ορισμού, και μετά ε, προβάλλατε αυτά τα στοιχεία Κάνατε προβολές με βάση αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι κάπως παράξενο από πλευράς επιστημονικής αυτό. Um, we had no other way. Δεν είχαμε άλλο τρόπο. Κάποιες χώρες από το δείγμα δεν είχαν εκτιμήσεις. Έπρεπε να τις κάνουμε βάση των πληροφοριών που είχαμε τις χώρες που μας έδωσαν πληροφορίες. Μετά εξετάζαμε 8 από τις 28 χώρες μας ανέθεσαν να δώσουμε κάποια εκτίμηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η προβολή αν ανωθεί έπρεπε να γίνει, αλλιώς δεν θα είχαμε βάση συγκρίσεως. Απάντηση. Αυτή η προβολή, αλλά οι οκτώ χώρε που ήταν η βάση για να βασιστείτε να κάνετε την προβολή, χρησιμοποιούσαν διαφορετικέ μεθοδολογίε και στη μελέτη ε, δεν ήταν διαφανέ ποιε μεθοδολογίε χρησιμοποιούσαν αυτέ οι χώρε, ούτω ώστε να καταλήξουν στοιχεία που σα δώσαν. Μπορείτε να μα δώσετε επίση για τις 8 αυτές χώρες τη μεθοδολογία που εφάρμοσαν οι χώρες για να καταλήξουν στα στοιχεία που σας έδωσαν. Γνέφει το μέρος του πάνελ, οπότε θα ανταλλάξουμε στοιχεία για την ανταλλαγή για την βάση δεδομένων. Ξέρουμε ότι υπάρχει έλλειψη εμπειρικών στοιχείων, χρησιμοποιούνται πολλές μεθοδολογίες. Αυτές ήταν επικρίσεις που ακούστηκαν και για τα κράτη-μέλη και δουλειά μας εδώ είναι να κλείσουμε το κενό όσον αφορά τα στοιχεία. Απευθύνθησαν εκκλήσει από το Κοινοβούλιο για κάτι τέτοιο. David Coburn του EFTD είναι επόμενος ομιλητής. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ίσως φρίξει ο κύριος Γκίγκολντ, αλλά συμφωνώ μαζί, μαζί του. Φρίτο κι εγώ λίγο. Δηλαδή οι μεθοδολογίες σας είναι τόσο αντιεπιστημονικές όπου είναι σαν να παίζουμε ε, ε, μακριά γαϊδούρα εδώ μέσα. Τέλος πάντων, κανείς δεν θέλει φοροδιαφυγή, αλλά πολλά άτομα και εταιρείε πρέπει να προστατεύσουν το χρήμα που βγάζουν σκληρά από σοσιαλιστικές κυβερνήσεις ε, ασταθείς ή αρπακτικές ή ανέντιμες. Οπότε περιγράψατε το Ηνωμένο Βασίλειο ως φορολογικό βασίλειο. Όχι. Είναι ένα ελκυστικό μέρος για τους επενδυτές με χαμηλούς φόρους που σέβεται την επιχειρηματική ελευθερία και τα χρήματα ατόμων ή εταιριών τα οποία βγάζουν εργαζόμενοι σκληρά. Δεν είναι ένα γραφειοκρατικό τέρας που ρουφάει τα χρήματα των φορολογουμένων για να πληρώσει τις μισθούς και τις συντάξεις των μεγαλοαστών στέλεχων της Ένωσης. Χαμηλή και δίκαιοι φόροι, κύριοι και κυρίες, θα μειώσουν την φοροαποφυγή. Ως επιχειρηματίας φρίτο από αυτή την, το, το μανιφέστο γραφειοκρατίας που παρουσιάζεται. Χρειαζόμαστε Brexit και μάλιστα σκληρό και μάλιστα τώρα. Φρίτο, πραγματικά υποτίθεται ότι θα έχουμε μια κοινή αγορά. Υποτίθεται ότι θα είχαμε ελεύθερο εμπόριο. Αυτό ήταν όλο. Εμείς δεν ζητήσαμε να κοιτάνε τους λογαριασμούς των ανθρώπων κάτι γραφειοκράτες. Δεν είναι βρετανικό αυτό και ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλες χώρες την πορεία προς την έξοδο. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας σχόλια για τον ευρωπαϊκό σοσιαλισμό και δεύτερον ε, δεν ξέρω αν διαβάσατε τη μελέτη αλλά τέλος πάντων νομίζω θα ήθελαν οι ερευνητέ να απαντήσουν δύο πράγματα δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα προσπαθήστε θέλετε ιδιωτικά ε, δηλαδή να λέτε ότι είναι γελία η μεθοδολογία μας δεν είναι σωστό Τι άλλη εναλλακτική είχαμε, απλά ρωτάμε. Και ζητάμε στοιχεία. Δεν υπάρχει εναλλακτικό τρόπος. Χρησιμοποιήσαμε ε, ένα εναλλακτικό μοντέλο. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εναλλακτικό μοντέλο, δηλαδή να μην μιλάμε με κανέναν. Αλλά νομίζω ότι το να ερχόμαστε σε επαφή με τις αρχές των κρατών μελών και να ζητάμε πληροφορίες, ε, εμένα μου φαίνεται ο μόνος τρόπος. Δεν είπαμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι φορολογικός παράδεισος. Είπαμε ότι κάποιοι το περιγράφουν ως τέτοιο, κάποιοι άλλοι όχι εμείς. Αυτή είναι η απάντησή μου. Για τα υπόλοιπα, όπω είπα, δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα άλλο. Μάλιστα, να προσθέσω ότι μέρος ε, των δηλώσεων αφορούσε τον κίνδυνο χρηματοδότησης Ισλαμικής τρομοκρατίας και νομίζω ότι και οι Βρετανοί πολίτες θα ενδιαφέρονταν για κάτι τέτοιο. Συμφωνείτε. Να, να πω ότι δεν θα παίξει καμία διαφορά. Αυτό γίνεται εδώ και αιώνες. Ε, πρόκειται για δικαιολογία για να χώνετε τη μύτη σας ε, και να χώνεστε εκεί που δεν σας παίρνουν. Η χρεοκοπημένη Ευρώπη και τα χρεοκοπημένα σοσιαλιστικά κράτη προσπαθούν να αρπάξουν περισσότερα λεφτά. Αυτό είναι όλο, έτσι, ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχει σχέση τώρα με την τρομοκρατία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης. Τα υπόλοιπα είναι μπουρδες. Δεν έχουμε κάποιον από το ΙΕΝΕΦ, e σωστά, καλά τα λέω. Δεν ακούω κάποια διαμαρτυρία, περνάμε στην Ρομπέρτα Μετσόλα του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τους ερευνητές για το έργο τους που ανάλυσαν τις επιδόσεις και τις επιδόσεις των χωρών που προσπαθούν να καταπολεμήσουν τα φαινόμενα φοροδιαφυγής, φοροποφυγής κτλ. Κοιτάξτε, αυτό που προσπαθεί να κάνει η Επιτροπή αυτή και τα αποτελέσματα στα οποία θα καταλήξει θα είναι συστάσεις ώστε η Ευρώπη να μην βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με μια τέτοια κατάσταση παράλυσης που διαπίστωσα και στη χώρα μου κι αλλού. Εγώ είμαι από την ε, Μάλτα και το λέω με βαριά καρδιά το τι έγινε την τελευταία εβδομάδα στη Μάλτα. Θα σας πω και μετά θα κάνω κάποιες ερωτήσεις που ελπίζω να προσπαθήσετε να μου απαντήσετε. Λοιπόν, γιατί είμαστε εδώ. Τα Panama papers έδειξαν ότι υπάρχει διαφθορά, υπάρχει φόρο διαφυγή, ακόμα και σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Στη δικιά μου κυβέρνηση της χώρας μου, δηλαδή τη σοσιαλιστιακή, έγιναν τέτοιες αποκαλύψεις που έδειξαν ότι ο τέος υπουργό μας ενέργειας και ο επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού είχαν μυστικές οικονομικές υπηρεσίες σε δικαιοδοσίες όπως είναι ο Παναμάς και η Παρθένη Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν τα μέσα στην Μάλτα δημοσίευσαν υπόνοιες ότι ο Πρωθυπουργό ή η γυναίκα του επίσης είχαν τέτοια ε, δομές στον Παναμά. Και επίσης ότι πήραν εκατομμύρια από εταιρείε που, είναι, που ανήκουν στην οικογένεια που κυβερνάει στο Αζερβαϊτζάν. Και πέρα από αυτά, ακόμα χειρότερα, και εδώ έρχομαι σε αυτό που συζητάμε σήμερα, η αστυνομία μέχρι τώρα αρνήθηκε ακόμα και να ασχοληθεί με την ιδέα της εξέτασης τέτοιων ισχυρισμών που έχουν να κάνουν με άτομα πολιτικά που έχουν εκτεθεί σε αυτού του είδους τις δομές. Ο επικεφαλής της αστυνομίας εξαλωρίζεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και είναι ο πέμπτος που έχουμε τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Και για να σας δώσω μια ιδέα για την έκταση της θεσμική κρίσης, σήμερα το πρωί η εθνική μας εφημερίδα λέει ότι πριν από ένα χρόνο η ομάδα έρευνας του ξεπλήματος χρήματος στην Μάλτα σύστησε στην αστυνομία να αναλάβει δράση κατά του επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού και η αστυνομία δεν το έκανε. Και η αστυνομία για προφανείς λόγους δεν πρόκειται να ενημερώσει την Europol και να τη ζητήσει να κάνει έρευνες. Αυτό όμως πονάει, ιδίως όταν η χώρα μου προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το εξάμεινο. Και θα ολοκληρώσω με μερικές ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στην απάντησή σας στον συνάδελφο Φαντεκάν λέγοντας του πώς μπορούμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα να έχει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός τη δυνατότητα να ερευνήσει χωρίς τη συνεργασία της χώρας μέλους. Τι γίνεται επίσης στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές ε, χώρες Στο κάτω-κάτω γιατί δημιουργήθηκε αυτή η Επιτροπή. Γιατί ο κόσμος θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει αυτό που οι χώρες μέλη από μόνες τους δεν μπόρεσαν να πετύχουν, δηλαδή να προστατεύσουν τον κόσμο από τέτοια σκάνδαλα. Απαντήσεις λοιπόν. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όσον αφορά τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις έρευνες δεν είναι ακριβώς μέσα στη μελέτη μας. Αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο της μελέτης μας. Αλλά υπάρχουν ε, βέβαια συστάσεις για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μπορούν να κάνουν οι μονάδες οικονομικών πληροφοριών, για διευθύνσεις οικονομικής αστυνομίας ουσιαστικά. Μιλάμε επίση για την υπηρεσία του Ευρωπαίου Συγγελέα Οικονομικού Εγκλήματο. που μπορεί να ασχοληθεί με τέτοια θέματα φοροδιαφυγής. Ίσως αυτό να είναι το κατάλληλο μέτρο για να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή. Αυτό θα μπορούσε να γίνει δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Στο Catch the Eye δεν βλέπω να υπάρχει καμιά ερώτηση. Ωραία. Τα καταφέραμε να είμαστε στην ώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις ερευνητές. Σίγουρα θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη βάση δεδομένων. Σας ευχαριστούμε για το έργο σας. Από εδώ και πέρα δικιά μας δουλειά είναι τα δικά σας συμπεράσματα να τα μεταφέρουμε στην δράση μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο χωρών μερών. Και στο δεύτερο πάνελ θα δούμε ακριβώ αυτά τα θέματα που ανέφερε και η συνάδελφος Ματσόλα, δηλαδή τι δράση έχουν αναλάβει μέχρι τώρα οι χώρε μέλη. Ευχαριστούμε. Um, λοιπόν, ενώ συμμαζεύονται και ετοιμάζονται οι ομιλητέ, πάμε στο δεύτερο πάνελ. Ευθύνε των κρατών τη της Ευρωπαϊκής Ενώσης για εφαρμοστέο δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποια είναι τα νομικά κενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, for, uh, preliminary... Προκατακτική επισκόπηση των επιδόσεων των αρμοδίων διοικητικών και δικαστικών αρχών σχετικά με τη φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Δεύτερη παρουσίαση. Προκαταρτική ανάλυση των επιδόσεων των αρμοδίων διοικητικών και δικαστικών αρχών όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και ξέπλυμα χρήματων. Σχολίασα ήδη την έλλειψη στοιχείων στα διάφορα κάτι μέλη και κάποια συνάδελφος ε, αναφέρθηκε σε αυτό, ο κ. Κάζα, και ήθελε να απαντήσει, αλλά πρέπει να προλάβει το αεροπλάνο του και έφυγε και δεν μπορούσαμε να τον έχουμε εδώ για να ακούσει τις απαντήσεις που θα δοθούν. Η έρευνα βασίζεται επί απαντήσεων κρατών μελών σε ερωτηματολόγιο που εξεδόθη από τον Πρόεδρο από του αρμόδιου υπουργού των κρατών μελών. Ζητήσαμε πληροφορίες για, τις εθνικού για ε, ορισμούς για τους τα φορολογικά δικήματα, τη σχέση μεταξύ φορολογικών ε, αρχών και μεθόδους εργασίας και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από αφορά μέτρα. Οι εθνικές συνεισφορές που λάβαμε έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΑ υπό τον τίτλο «Έτοιμα για συνεισφορά από, από κρατών μελών». Καλώ τους ομιλητές να πάρουν το λόγο. Κυρία Σέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Στέφαν Ρέγο ζητήσει συγγνώμη που ήταν υπεύθυνο για τη μελέτη. Αλλά περιμένει να γεννήσει η γυναίκα του και δεν μπορεί να είναι εδώ. Πολύ σωστός λόγος και συγχαρητήρια στην γυναίκα του. Θα παρουσιάσουμε ποια είναι η κατάσταση. Μέσω της μελέτης θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, η Ελοντή και εγώ, να απαντήσουμε. Θα διαβιβάσουμε και τυχόν ερωτήσεις στον Στεφάν για να απαντήσει αργότερα, στο, να απαντώντας τον καθέναν από εσά λεπτομερέστερα. Ποια είναι η κατάσταση, λοιπόν, για τη μελέτη. Αυτή η δημοσίευση θα είναι ανάλυση. Συντάσσεται από την αξιολόγηση εκ των υστέρων του EPRS, εφαρμογή δράσεων. Αναλύουμε τα συστήματα και τις δυνατότητες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, των απατών και του ξεπλήματος χρήματος. Ε, προστευμένος ε, προσωρινός τίτλο είναι Οι επιδόσει των κατώμενων τη Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν τη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, απάτη στον τομέα των φόρων και ξέπλυμα χρήματο. Στόχο 7 Ιουλίου να δημοσιευτεί φέτο το έγγραφο στο τέλο λοιπόν, τη περίοδου. Βασιζόμαστε σε απαντήσει ερωτηματολογίου ο πρόεδρος Επιτροπή Έρευνα, ο Δ. Λάγκεν, έστειλε το ερωτηματολόγιο στους Υπουργού Οικονομικών και Δικαιοσύνη των κρατών της Ευρωπαϊκή Ενώσεω στι 23 Νοεμβρίου του 2016. Λοιπόν, μερικά λόγια να πω τώρα όσον αφορά τα μέλη τη ομάδα μα. Δημιουργήθηκε αυτή η ιστορική ομάδα μελέτη έρευνα. Ο Στέφαν Ρέινολτζ είναι υπεύθυνο για τη βασική ανάλυση και τη σύνταξη του κειμένου. Επίση, περιλαμβάνει ομάδα άλλου τρει αναλυτέ εκ των υστέρων. Πέραν από τον Στεφάν έχουμε την Ελοντή Τυριούν, η οποία θα μιλήσει αργότερα μετά από μένα, που εστιάζεται επί της συγκριτικής νομικής μελέτης των εθνικών ορισμών, των εθνικών νόμων και των εφαρμοστικών διατάξεων που σχετίζονται με φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Εγώ θα μιλήσω για τα στοιχεία της αναλύσεως που αφορούν τις μονάδες συλλογής στοιχείων για τα χρηματοστατικά, και να δούμε κατά πόσο ταιριάζει η ενδελεχή ανάλυση με αυτά τα στοιχεία και πόσο τα στοιχεία αυτά θα ταιριάζουν και με την έκθεση που θα παρουσιάσουμε τελικά. Η ομάδα επίση επικουρείται από τη συνάδελφο Μωρή Χάμελερς που αναλύει τα στατιστικά στοιχεία των κρατών μελών και τέλο το έγγραφο θα αποσταλεί επισήμω εξωτερικό αναλυτή και εξεταστή την καθηγήτρια Μπριγκίτα Ούγκαρ που συναντήσατε σε άλλη ακρόαση από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτη. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τώρα τις ερωτήσεις που στείλαμε στα κράτη-μέλη. Να το ερωτηματολόγιο. Γενικά λοιπόν το ερωτηματολόγιο ζητούσε λεπτομέρειες. Να μας δώσει τα κράτη-μέλη τους νομικούς ορισμούς των αδικημάτων σχετικών φορολογικά και το πλήρες ε, όσον αφορά τα ενδιαφέροντα του ΠΑΝΑ. Οι λεπτομέρειες των εργασιών των αρχών όσον αφορά τις ύποπτες συναλλαγές και το πώς ε, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συντώνησαν τις εργασίε του. Το ερωτηματολόγιο επίσης συμπεριλάμβανε πληροφορίες που ζητούσαμε για εφαρμοστέο και εφαρμόσιμο καθεστώς για κυρώσεις και διώξεις για τα αδικήματα τα φορολογικά. Ζητούσαμε λεπτομέρειες για τα είδη των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν, λεπτομέρειες δραστηριότητε των εθνικών εποπτικών αρχών για τα οικονομικά και ιδιαίτερα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τα είδη των εμπλεκομένων εταιριών, τις κυρώσει για τα δικήματα και τα πρόστιμα. Τέλος, το ερωτηματολόγιο ζητούσε να περιγραφεί κατάσταση όσον αφορά τις έρευνες των κρατών μελών που σχετίζονται με τα έγγραφα του Παναμά και τις διαρροές ε, των Μπαχάμας. Ε, τώρα, όσον αφορά τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, κάναμε μια ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, η οποία θα εδράζεται βασικά επί των πληροφοριών που μας έδωσαν τα κράτη-μέλη ε, απαντώντας στο ερωτηματολόγιο. Πέραν αυτού, ε, πληροφορίες που περιέχονται σε επίσημες εκθέσεις των κρατών μελών, αιτήσεις εκθέσεις συνήθω, που ε, αναφέρονται εδώ, επίσης αξιολογούνται και βεβαίως θα ληφθούν υπόψη στη μελέτη μας. Λοιπόν, αυτές είναι οι ερωτήσεις που θέσαμε και οι απαντήσεις των κρατών μελών. Είναι δημόσια όλα αυτά. Μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά στην ιστοσελίδα Πανά. Βλέπετε εξάλλου και την ιστοσελίδα στην οθόνη. Έτσι λοιπόν παρουσιάζεται η ιστοσελίδα μας. Ως υπενθύμηση, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα κράτη-μέλη απαντήσεις και να ακολουθήσουν τη σειρά των ερωτήσεων. Ο Πρόεδρος επίσης ζήτησε οι μασικέ πληροφορίες να ταιριάζουν με διάφορες ε, διασυνδέσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες σε παραρτήματα δεν υπήρχε όριο όσον αφορά τον όγκο πληροφοριών των παραρτημάτων. Προθεσμία ήταν 15 Ιανουαρίου 2017 που είχε τεθεί για όλα τα κράτη-μέλη να απαντήσουν μέχρι τότε. Η πρώτη παρατήρηση ποια είναι. Κανένα κάτω μέλος δεν συμμορφώθηκε εγκαίρως. Αυτό ίσως είναι κατανοητό, διότι όπως αναφέρθηκε προς τον Στέφαν Ρέινολντ σε ανεπίσημες επαφέ, η συλλογή των πληροφοριών που το ήταν κάτι μακροσκελές και δυσχερές ω εγχείρημα και η προθεσμία ήταν πολύ πρωίμη. Τότε η εντολή Πανά δεν είχε παραταθεί. Οπότε στο τέλος πέντε απαντήσεις παρελήθησαν τον μήνα Ιανουάριο, 13 τον μήνα Φεβρουάριο, άλλες τέσσερις κατέφθασαν τον μήνα Μάρτιο, δύο τον Απρίλιο και περιμένουμε, περιμένουμε άλλες τρεις τώρα. Από σήμερα λοιπόν η Ουγγαρία μας είπε ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ουγγαρίας, ε, τελεί υπό ε, υπηρεσιακές διαβουλεύσεις. Αλλά δεν μας είπαν πότε θα καταφάσει το έγγραφο. Η Ισπανία και η Δανία ακόμα δεν έδωσαν απάντηση. Παρόλο που μας το υποσχέθηκαν. Ούτε η Μάλτα. Και δεν έχουμε κανένα μαντάτο για το τι κάνει η Μάλτα. Εν πάση περιπτώσει. κλείνοντα λοιπόν, όσο αυτή τη διαφάνεια. Με το σταγονόμετρο έρχονται πληροφορίε από τα κάτι μέλη και πάντα κυνηγάμε με το δίκανο και γι' αυτό έχουμε καθυστερήσει εμεί και δεν έχουμε μπορέσει να δημοσιεύσουμε το έγγραφο το Μάρτιο όπω προβλεπόταν. Όμω, έχουμε ημερομηνία 7 Ιουλίου τώρα για δημοσίευση. Άρα μπορούμε τελικά να λάβουμε τι πληροφορίε και να τι αναλύσουμε. Έχουμε καιρό. Και οι ευρωβουλευτέ μπορούν να εξετάσουν τα πορίσματα πριν την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στο σχέδιο εκθέσεω που έχει καθοριστεί για 5 Σεπτεμβρίου του έτου 2017. Λοιπόν, από την προκατατική ανάλυση των στοιχείων των κρατών μελών, τι βλέπουμε, τα κράτη-μέλη μπορούν ε, να πούμε ότι οι απαντήσεις που δώσαμε μπαίνουν σε τρεις κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα, ελάχιστες απαντήσεις. Υπολείπονται των προσδοκιών αυτές. Δηλαδή λίγες μέχρι μηδέν στατιστικές πληροφορίες και ελάχιστη ανάλυση. Στο τέλος αυτό θα είναι περίπου το 1 τέταρτο των απαντήσεων. Λουξεμβούργο, Φερρυπίνα ανήκει σε αυτή την ομάδα του Λουξεμβούργου. Δεύτερον, εκτιμήσαμε ότι περισσότερες απαντήσεις αποτελούνται από ικανοποιητικές ε, απαντήσεις. Αυτές που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας θα οδηγήσουν σε κάποια χρήσιμα στοιχεία και αναλυτικά στοιχεία. Παρόλο που ξέρετε μας λείπουν κάποια πράγματα. Αυτή η ομάδα συμπεριλαμβάνει διάφορες χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης αλλά και τη Γερμανία τις οποίες η απάντηση αρχικά θεωρείται πάρα πολύ ποιοτική, αλλά ε, τελικά υπήρξε ασαφή σε κάποια σημεία. Εκεί συμπεριλαμβάνεται και το Ηνωμένο Βασίλειο, που ήταν πολύ καλό στα στοιχεία, αλλά έχει αδυναμίες, αδυναμίες όσον αφορά την περιγραφή του νομικού συστήματος. Τέλος, μικρότερος αριθμός ποιοτικών απαντήσεων, και εδώ έκλεισε και το μικρόφωνο. Α, συγγνώμη. Μικρότερος αριθμός ποιοτικών απαντήσεων, υπεράνω των προσδοκιών κατέφτασε. Εκεί όλε οι απαντήσει δίνονται λεπτομερώ ή περισσότερε. Η καλύτερη συνεισφορά κατά την άποψή μου είναι από την Ολλανδία, τη Σουηδία αλλά και τη Φιλανδία. Ποια είναι η γενική εντύπωση, ότι κάποια κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου Φερρυπίν, απάντησαν με αρκετά μεγάλο ενθουσιασμό στην απάντησή μα για πληροφορίε. Επίση, είναι σαφέ ότι μια άλλη ομάδα κρατών μελών και κάνουν το αντίθετο και απάντησαν με έναν τρόπο που απλώς είναι επαρκής θα έλεγα. Χωρίς να μας δώσουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Έκαναν τα ελάχιστα, εν πάση περιπτώσει. Αυτά που έχουμε θα επεξεργαστούμε, τι να κάνουμε. Και όπως θα εξηγήσω αργότερα, χρόνο επιτρέποντος, ίσως να υπάρχει δυνατότητα τα κράτη-μέλη να προσθέσουν κάποια στοιχεία ή τουλάχιστον να ελέγξουν ότι πράγματι τα στοιχεία τους είναι σωστά. Τέλος πάντων, Όσο έχουν τα πράγματα, το πρωτοτυπικό έργο μας αποκαλύπτει ότι η συγκριτική ανάλυση θα είναι περιπλοκότατη. Ποικίλουν οι απαντήσεις σημαντικά σε μορφή, σε μήκος, σε αριθμό περιεχόμενο παραρτημάτων, στο βαθμό των πληροφοριών που παρέχονται, στην προσβασιμότητα των πληροφοριών και πράγματι οι απαντήσεις δεν είναι πάντα γραπτές σαφώς και δεν είναι καν συνεκτικά κάποια στοιχεία. Και τώρα θα αφήσω την Ελοντή γου τη συνάδελφό μου, να παρουσιάσει τι αρχικέ μας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρουσιάσω τις αρχικές μας παρατηρήσεις και είμαστε στη διαδικασία ανάλυσης τώρα των εθνικών διατάξεων για την φόρο αποφυγή, την φόρο διαφυγή και την νομοποίηση παράνομων εσόδων και εξετάζουμε πώς αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις. Και θα εξετάσουμε επίσης και τους ε, στόχους, την, το είδος των παραβάσεων αυτών και τις διατάξεις που ισχύουν. Είχαμε απαντήσεις όσον αφορά την φοροποφυγή και το ξέπλυμα ε, την ομοποίηση παράνομου χρήματος από όλες τις χώρες και τι ισχύει για την νομοποίηση παράνομων εσόδων όλες οι χώρες το θεωρούν ότι είναι παράβαση. Υπάρχει ορισμός ο οποίος ε, διεθνώς συμπίπτει. Υπό το φως αυτό λοιπόν οι συστάσεις μας συνδέουν τα αποτελέσματα της ερευνάς μας και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, αποφυγή της νομοποίησης παράνομου χρήματος που είχαμε από το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Οι περισσότερες χώρες δίνουν κάποιες λεπτομέρειες επίσης και για την νομοθεσία τους όσον αφορά τη φοροαποφυγή. Μερικές χώρες όμως αναφέρονται μόνο στις γενικές νομικές τους πράξεις και όχι στις ειδικέ διατάξεις, πράγμα το οποίο μας έκανε πιο δύσκολη την ανάλυση από ό,τι είχαμε προβλέψει από την αρχή. Ε, βλέπουμε ότι οι χώρε μέλη διαθέτουν διαφορετικού νομικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση τη ε, φοροδιαφυγή και υπάρχει διάκριση ανάμεσα στις παραβάσεις. Για την φόρο αποφυγή, δεδομένου ότι η πρακτική αυτή την αντιλαμβανόμαστε όλοι σαν μια γκρίζα ζώνη, Λίγες χώρες έχουν ένα νομικό πλαίσιο προκειμένου να προχωρούν στη δίωξη κάποιου ο οποίος προς το συμφέρον του χρησιμοποιεί ε, τέτοιες ε, συμπεριφορές αποφυγής. Στην ανάλυση μας προσπαθούμε να εντοπίσουμε ένα μοντέλο, ένα πρότυπο που να ακολουθούν όλες οι χώρες για να καταλάβουμε καλύτερα και τα ποιοτικά και τα ποσοτικά στοιχεία που μας έδωσαν οι χώρες μέλη. Στις απαντήσεις τους όσον αφορά την διοικητική ικανότητα και τα, τις φορολογικές απάτες, όλες οι χώρες εξήγησαν πόσο συλλέγουν φόρους πρώτα απ' όλα, ποιος είναι ο μηχανισμός. Και ήδη εδώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών μελών και όσον αφορά την αναφορά των περιπτώσεων και όσον αφορά τον αριθμό των περιπτώσεων που έφτασαν στα δικαστήρια, τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και γενικά το, την αξία του ποσού το οποίο ανακτήθηκε. Επίσης εξηγούν τις δυνατότητες που έχουν οι διάφορες μονάδες τους που είναι οι διευθύνσεις οικονομικής αστυνομίας. Εξήγησαν όλες οι χώρες πώς αναλύουν οι μονάδες αυτές τα δεδομένα. Και επιπλέον οι χώρες μέλη ως επιτοπλίστων μας παρουσίασαν και κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις και εξήγησαν πώς οι μονάδες αυτές οικονομικής αστυνομίας συνεργάζονται ε, με άλλες αρχές για να ανταλλάξουν πληροφορίες. Παρατηρούμε επίσης πόσο μία ύποπτη συναλλαγή αναλύεται από τις μονάδες αυτές και πώς η πληροφορία αυτή στη συνέχεια πηγαίνει στην ε, αρχή στην οποία πρέπει να πάει ανάλογα βέβαια με το τι ήθιστε στην κάθε χώρα μέλος. Συνήθως τους εισαγγελείς ή στις φορολογικές αρχές προκειμένου να ερευνήσουν παρετέρω τις περιπτώσεις αυτές τις ύποπτες. Επίσης αναφέρουν πολλές πώς προχωράει η διαδικασία σε κυρώσεις ή σε παρετέρω δικαστικές διαδικασίες ή ακόμα και σε ποινικά δικαστήρια όταν πρόκειται βέβαια για πολύ μεγάλες φορολογικές απάτες και εγκλήματα. Αναφέρονται λοιπόν οι περιπτώσει που έχουν εξεταστεί από τι Διευθύνσει Οικονομική Αστυνομία αλλά και από του εισαγγελεί οικονομικών ε, εγκλημάτων με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Βέβαια, όχι από όλε τι χώρε. Οπότε και εδώ υπάρχουν ε, όρια στη συγκρισιμότητα των στοιχείων. Άρα και στην ανάλυση μας. Πάντως έχουμε αρκετά στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν τώρα να πούμε ότι η φοροαποφυγή, η μη πληρωμή ΦΠΑ οδηγούν σε σημαντικές επιπτώσεις. Υπάρχουν ε, βέβαια περιορισμοί στις χώρες μέλη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις φορολογικές απάτες. Έχουν εξηγήσει πολλές χώρες επίσης τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοιες φορολογικές απάτες όταν αυτές είναι διεθνείς ή διασυνοριακές έχουν εκφράσει και δυσκολίες για την αντιμετώπιση των ε, εγκληματικών οργανώσεων. Πολύ συχνά πρέπει να δούμε μήπως τελικά για να αντιμετωπιστούν κάποιες περιπτώσεις πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει κάποια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση γιατί έχουν ε, έτσι κι αλλιώς διασυνοριακή διάσταση βάσει των στοιχείων που έχουμε, ε, κάποιες φορολογικές απάτες έχουν να κάνουν έτσι κι αλλιώς με εγκληματικές οργανώσεις και γι' αυτό χρειάζεται να ασχοληθεί με αυτό ο Ευρωπαίος εισαγγελέα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα της σημερινής συζήτησης. Επίσης, έχουμε προχωρήσει σε ανάλυση αρκετά πλήρη αλλά και πάλι κάποια από τις πληροφορίες που μας έχουν ε, έρθει είναι κάτω από τις προσδοκίες μας. Φαίνεται πάντως έτσι καλλιώς ότι υπάρχουν διαφορές στις ε, διαδικασίες που ακολουθούν οι διάφορες χώρες και τη στρατηγική τους τόσο όσον αφορά την φορολογία αλλά όσο και την επίτευξη των φορολογικών στόχων. Από τη μια διαπιστεύουμε ότι υπάρχουν ε, συστήματα τα οποία επιβάλλουν περισσότερες κυρώσεις, είναι πιο αυστηρά για να οδηγήσουν στην αποτροπή από τέτοιε φορολογικές παραβιάσεις. Από την άλλη μεριά υπάρχουν συστήματα τα οποία προσπαθούν να ενθερίνουν τη συμμόρφωση. Υπάρχει και διαφορά ανάμεσα στις χώρες μέλη όπου έχουν ευνοϊκές φορολογικές πολιτικές βάσει του αναπτυξιακού μοντέλου και εκείνες οι χώρες που έχουν λιγότερο ευνοϊκά φορολογικά συστήματα. Επίσης, το θέμα του ελέγχου και της διαφάνειας διαφέρει από χώρα σε χώρα και έχει να κάνει πιο πολύ με τη διοικητική νοοτροπία που επικρατεί. Στις βόρειες χώρες, στην Ευρώπη, δίνουν περισσότερους πόρους για να έχουν εθνικές εκθέσεις ή και αιτήσεις εκθέσεις δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τα φορολογικά και τις εγκληματικές πρακτικές σε βάρος των φορολογικών εσόδων με διαφάνεια. Άλλες πάλι τέτοιες ε, εκθέσεις δεν τις δημοσιεύουν. Οι χώρες μέλη έχουν απαντήσει επίσης διαφορετικά στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα Panama Papers και Bahama Leaks. Δεν ε, αναγνωρίζονται πάντα, κυρίως στις χώρες εκείνες που έχουν πιο νομικήστική αντίδραση και δεν υπάρχει πάντα επαρκής επικοινωνία όσον αφορά τις πληροφορίες και αυτό συμβαίνει στις περισσότερες χώρες. Κάποιες χώρες συνεχίζουν την ανάλυση των δύο αυτών περιπτώσεων. Οι χώρες μέλη Απάντησαν πάντως με λεπτομέρειες όσον αφορά τις πρωτοβουλίες τους προκειμένου να αναλύσουν το τι έχει γίνει στις χώρες αυτές με τα Panama Papers και δίνουν στατιστικά στοιχεία. Κάποιες άλλες λιγότερο. Όσον αφορά τώρα τις δράσεις που έχουν αναλάβει οι χώρες μετά τα Panama Papers, το Ηνωμένο Βασίλειο και κάτω χώρες έδωσαν περισσότερες πληροφορίες, όπως επίσης και η Γερμανία, ενώ άλλες δεν έδωσαν αρκετά στοιχεία, σχεδόν τίποτα. Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, πολύ συχνά διαβάσαμε ότι α, είναι πολύ νωρίς για να σας πούμε περισσότερα. Δεύτερον, κάποιες χώρες λένε ότι έχουν ήδη αρκετές περιπτώσεις στα Panama Papers που εξετάζουν και ότι τα εξετάζαν ήδη, εξετάζαν ήδη αυτές τις περιπτώσεις και τα Panama Papers το μόνο που κάνανε είναι ότι τους επιβεβαίωσαν τις υποψίες. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει δυσκολία να ε, φτάσει κανείς στην πληροφορία του Διεθνούς Ομίλου Reporters. Άλλες χώρες είπαν ότι τα Bahamas Leaks, αντίθεση με τα Panama Papers, ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν γιατί το υλικό είναι πολύ φτωχό. Τέλος, δεν μπορώ να σας πω ακόμα κατά πόσο οι περισσότερες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με τα Panama Papers έχουν να κάνουν περισσότερο με ατομικές περιπτώσεις ή με εταιρείε. Είναι κάτι πάντως που εξετάζεται. Τώρα για να βοηθήσουμε στο αναλυτικό έργο, επειδή ακριβώς και η δομή και το περιεχόμενο είναι εντελώ διαφορετικό στις πληροφορίες που πήραμε από τι χώρε μέλη, προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε το βασικό μήνυμα και τα βασικά στοιχεία τα οποία πήραμε. Τώρα αναλύουμε με ένα ε, φάκελο αναχώρα μέλος, με ένα δελτίο, συγκεντρώνοντας εκεί τις πληροφορίες που έχουμε πάρει και προσπαθώντας να τις απλοποιήσουμε. Αυτή η εικόνα είναι ένα παράδειγμα για τη Φιλανδία. Οι πληροφορίες που αναφέρονται εδώ βασίζονται στις πληροφορίες που μας έδωσε το συγκεκριμένο ε, κράτος μέλο με ό,τι παρατήματα και πληροφορίες μας έχει στείλει. Για να καλύψουμε τα κενά ή οποιαδήποτε λάθη στην μεταγραφή, το δελτίο αυτό θα πάει στις αρμόδιες αρχές της χώρας μέλους για να σχολιάσει. Αυτό δίνει και την ευκαιρία στις χώρες μέλη να συμπληρώσουν με πληροφορίες τα δελτία αυτά. Αφού λοιπόν συμπληρώσουν με σχόλια το δελτίο αυτό οι χώρες μέλη, θα έχουμε και άλλε, άλλους ποιοτικού ελέγχους. Πρώτον, οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εξετάσουν άτυπα τα δελτία αυτά για να δουν αν, μπορούμε, αν μπορούν να προσθέσουν κάτι στην ανάλυση μας. Και δεύτερον, όπως είπε και η συνάδελφος πριν, θα έχουμε και μία peer review αναθεώρηση από τους ομολόγους από τη Σχολή Οικονομικών της Ουτρέχτης που έκανε το σχέδιο το 2013 για την αποτελεσματικότητα, την οικονομική και νομική και για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις, τα εγκλήματα, τα οικονομικά. Θα μας βοηθήσουν λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη και δραστηριότητες offshore. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ό,τι ερωτήσεις έχετε θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Thank you very much indeed and... Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ και βεβαίω ε, να μεταφέρετε τις ευχές μου στον συναδελφό σας ε, και την οικογένειά του. Περνάμε στην επόμενη παρουσίαση και μετά θα έχουμε ένα τελευταίο γύρο ομιλητών. Κύριε Μιτσέλο, είστε από το Διεθνές Κέντρο Συγκριτικής Εκκληματολογίας από το Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ στον Καναδά και θα μας παρουσιάσει μια μελέτη η οποία αφορά την συνεργασία για την καταπολέμηση του φορολογικού εγκλήματος. Βασίζεται λοιπόν σε χαρτογράφηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνει μια συγκριτική ανάλυση για τις μονάδες πληροφοριών και εστιάζει μετά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές. να το δείγμα και δύο κράτη-μέλη τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μια τέτοια μονάδα από ευρωπαϊκή χώρα, την Ελβετία, μεγάλο οικονομικό κέντρο, και τον Καναδά. Και στόχο έχει να προσφέρει μια καλύτερη αντίληψη ε, του τι συμβαίνει με τις αρμοδιότητες των μονάδων συλλογής πληροφοριών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Δίνω λοιπόν τον λόγο στον δόκτωρα Αμιτσέλο για... Α, λάθος. Εσείς, εσείς ξεκινάτε. Κυρία Σέιρα, λοιπόν, και μετά ο κύριος Αμιτσέλη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. είναι στην υπηρεσία έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν αιτήματος επιτροπής που μια μελέτη για τις μονάδες ε, δημοσιονομικών πληροφοριών. Η μελέτη μας, όπως ξέρετε, ξεκίνησε τον Μάρτιο και είχε δύο μέρη. Μία ανάλυση για τις μονάδες ε, οικονομικών πληροφοριών και το νομικό πλαίσιο της Ένωσης και μία συγκριτική ανάλυση τεσσάρων συγκεκριμένων τέτοιων ομάδων. Γαλλία, σε, είπα, σε, με συγχωρείτε, Βασίλειο, Γαλλία, Καναδά και Ελβετία. Να σα τι είναι η μονάδα οικονομικών πληροφοριών. Πρόκειται συνήθω για μια εθνική υπηρεσία με στόχο την συλλογή, ανάλυση και διάδοση οικονομικών πληροφοριών για να, ξεπληθεί το ξε... για να καταπολεμηθεί το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της δρομοκρατίας. Λαμβάνουν λοιπόν εκθέσεις ύποπτων συναλλαγών που στέλνουν διάφοροι φορείς οι οποίοι σύμφωνα με την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λογιστές, ε, φοροτεχνικοί, κτηματομεσίτες και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Όλοι αυτοί πρέπει να σέβονται και να, τον νόμο και να ενημερώσουν τις αρμόδιες μονάδες ε, εάν θεωρούν ότι υπάρχει απόπειρα ξεπλήματος χρήματος και οι μονάδες αυτές αναλύουν τις σχετικές πληροφορίες και αν τους μεταδίδουν για περαιτέρω έρευνα όσον αφορά λοιπόν το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα αναφερθώ στην κατάσταση που υπάρχει και στην καταγραφή που κάναμε για την πλατφόρμα η οποία είναι η πλατφόρμα την οποία συντονίζει η Κομισιόν για να διευκολύνει τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών Όσον αφορά λοιπόν την καταπολέμηση των φορολογικών εγκλημάτων, η ανάλυση μας ε, οδήγησε στο να βρούμε τρεις κυρίες προκλήσεις. Πρώτα απ' όλα στο εθνικό επίπεδο η συνεργασία μεταξύ των μονάδων πληροφοριών και των φορολογικών αρχών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Και υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωση. Θα μπορούσαν να γίνουν κάποια εθνικά μνημόνια συναντήληψης μεταξύ των υπηρεσιών αυτών για να μην γίνεται δύο φορές η ίδια δουλειά και να βελτιωθεί η αμοιβαία γνωμοσύνη. Δεύτερον, η έλλειψη εθνικών βάσεων δεδομένων για τους κατόχους τραπεζικών λογαριασμών και των πραγματικών ιδιοκτητών είναι ένας τομέας ανησυχίας. Ε, κεντρικά αρχεία ναι, ε, τέτοια κατόχων τραπεζικών λογαριασμών δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Και βεβαίως η τέταρτη οδηγία συνιστά στα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είναι υποχρέωση. Η υποχρέωση δε για κεντρικά τέτοια αρχεία δεν έχει ε, μέχρι σήμερα εκπληρωθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη έχουν ακόμα τρει μήνες για να μεταφέρουν αυτές τι διατάξεις. Τρίτον, όσον αφορά την συνεργασία μεταξύ των μονάδων πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι διαφορές ε, όσον αφορά τις αξιόπινες πράξεις συχνά αποτελούν εμπόδιο στην ανταλλαγή πληροφοριών. Πράγματι, η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί αντικείμενο άρνησης όταν μια αξιόπινη πράξη δεν τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο σε άλλη χώρα. Και αυτό σημαίνει πολύ συχνά σε φορολογικά αισθήματα. Παρά τις προκλήσεις αυτές πρέπει να σημειώσουμε πως κάποιες διατάξεις της οδηγίας ε, κατά του ξεπλήματος χρήματος που πρέπει να μεταφέρθει στην νομοθεσία φέτος τον Ιούνιο αφορούν την βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης. Δηλαδή έχει στόχο να βελτιώσει την καθυστέρηση και να δώσει την δυνατότητα μονάδες πληροφοριών να έρθουν πρώτε σε επαφή για, με τις τράπεζες για τέτοιες πληροφορίες και ξεκαθαρίζει επίσης τις διαφορές μεταξύ των ορισμών στην ομοθεσία των αξιόπινων φορολογικών πράξεων και το ότι δεν θα εμποδίζουν αυτές την μετάδοση πληροφοριών. Λέει ότι οι μονάδες πληροφοριών θα πρέπει να μεταδίδουν τις πληροφορίες εάν είναι αξιόπινη η πράξη στην άλλη χώρα. Επιπλέον, οι μονάδε πληροφοριών θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλες τις εθνικές αρμοδιότητες για να απαντήσουν σε κάποιο αίτημα. Οπότε, απομένει βέβαια να δούμε αν θα εφαρμοστούν και θα μεταφερθούν σωστά στο εθνικό δίκαιο αυτές οι διατάξει. Όσον αφορά το γενικό πλαίσιο της Ένωσης, πρέπει να σημειώσουμε και καταλήγω εδώ ότι η Κομισιόν έχει υποβάλει μια πρόταση οδηγία τον Δεκέμβριο με στόχο να ενισχύσει την εναρμόνιση του ορισμού του ξεπλήματος χρήματος και των σχετικών πράξεων. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Δ. Αντώνια Μισελ για να μας παρουσιάσει τα ευρήματα της ανάλυσης που έκανε στις τέσσερις χώρες και θα μας πει τις αρμοδιότητες των άλλων πληροφοριών και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαρά που είμαι σήμερα να παρουσιάσω αυτή την έρευνα μετά την δύσκολη νυχτερινή μου πτήση. Χάρηκα που κατέθασα για να παρουσιάσω την έρευνά. Την έκανα με δύο συναδέλφους. για τον ε, ρόλο που διαματίζεται από τους φορείς καταπολέμησης των φορολογικών εγκλημάτων με την εφαρμογή τριών οδηγιών και την καταπολέμηση ξεπλήματος χρήματος. Πρώτο, σύντομη ιστορική επισκόπηση. Να καταλάβουμε το ρόλο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μονάδες συλλογής πληροφοριών για το οικονομικό έγκλημα. Λοιπόν, οι μονάδες καταπολεμήσεις του οικονομικού εγκλήματος είναι οι βασικοί εθνικοί θεσμοί που καταπολεμούν το ξέπλυμα χρήματος. Θέλουμε να καταλάβουμε το ρόλο τους, τις πρακτικές που ακολουθούν, το διακύβευμα και γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούμε με το βρώμικο χρήμα. Από την πρώτη οδηγία του 1991 μέχρι την τελευταία, που έγινε πριν από μερικά χρόνια, τι βλέπουμε όσον αφορά το βρώμικο χρήμα. Άλλαξε η έννοια. Στην πρώτη οδηγία το βρώμικο χρήμα ήταν συνώνυμο του χρήματος για τα, από τα ναρκωτικά. Και τώρα σχετίζεται με κάθε μορφή εγκληματικών οικονομικών ροών, παρανόμων, από ναρκωτικά τρομοκρατική χρηματοδότηση τρομοκρατών, διαφθορά, φοροαποφυγή κλπ. Και, το καθεξής. και αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο όσον αφορά τη λογική, το ρόλο και την ταυτότητα της μονάδας κατά πολεμής του οικονομικού εγκλήματος. Όπως γνωρίζετε, το ξέπλυμα χρήματος μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα εξαρτώμενο αδίκημα. Εξαρτάται από πρώτερο έγκλημα, από το οποίο προήλθε το χρήμα που ξεπλένεται. Γι' αυτό είναι και βρώμικο. Όπως ανέφερα αρχικά, αυτές οι μονάδες καταπολεμήσεως του οικονομικού εγκλήματος σχεδιάστηκαν να καταπολεμήσουν αυτά τα έσοδα από το έγκλημα σχετικά τα ναρκωτικά και τώρα παρουσιάζονται σαν βασικός κόμβος συλλογή πληροφοριών σχετικά με όλα αυτά τα δικήματα. Κάθε μορφή οικονομικού εγκλήματος. Μεγάλη διαφορά σε σχέση με την αρχή. Οπότε τώρα που συμπεριλήφθη ρητά η φόρα αποφυγή στο πλαίσιο, αυτό είναι σημαντικότατα έλεγε. Ιστορικός πως από την αρχή της δεκαετίας του 90 υπήρχε ε, αποκλεισμός εξαίρεση των φορολογικών θεμάτων και είχε ερμηνευθεί σαν ε, θετική ανοχή εναντί των σχετικών εγκληματιών. Τώρα το φορολογικό έγκλημα έγινε προηγούμενο έγκλημα για το ξέπλυμα του χρήματος και τέθη τέρμα στην επιλεκτική ανοχή. Δεύτερη αλλαγή. Και αλλαγή νοοτροπία όσον αφορά το έργο των μονάδων αυτών ποιο είναι. Συμπερίληψη φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής τροποποιεί τη λογική που ακολουθούν οι μονάδες. Κανονικά οι μονάδες αυτές παρακολουθούν την παράνομη προέλευση του χρήματος. Όσον αφορά τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή είναι διαφορετικά τα πράγματα λίγο. Διότι η προέλευση των χρημάτων μπορεί να είναι παράνομη, αλλά ο τρόπο που χρησιμοποιείται για φοροαποφυγή ε, μπορεί να το κάνει παράνομο. Ίσως ο προορισμό και όχι η προέλευση να κάνει τη διαφορά. Εστιάζεσαι λοιπόν και στην προέλευση τώρα, αλλά και στον προορισμό και τη χρήση. Άλλαξε λοιπόν η προσέγγιση άλλαξε αυτό πριν συμπεριλάβουμε τη φοροδιαφυγή. Αλλά άλλαξε το 2001 όταν θέλαμε να αντιμετωπίσουμε τη χρηματοδότηση τρομοκρατών. Η χρηματοδότηση των τρομοκρατών, τι αντίκτυπο είχε. Η συμπερίληψη της χρηματοδότησης είχε τεράστιο αντίκτυπο όσον αφορά τον όλο μηχανισμό καταπολεμήσεως του ξεπλήματος χρήματος. Όσον αφορά το τομέα καταπολεμής οικονομικού εγκλήματος γενικότερα, συζητείται το θέμα. Κάποιοι λένε ότι εν ονόματι χρηματοδότηση τρομοκρατών οι μονάδες καταπολεμήσεως εγκλήματος παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα οικονομικά, εξουσίες, ανθρώπους, προσωπικό. Άρα έχουμε συνέπειες μόχλευσης στην προσπάθεια καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος. Άρα η καταπολέμηση χρηματοδότησης τρομοκρατών είναι κάτι χρήσιμο για κάθε μορφή οικονομικού εγκλήματο. Κάποιοι ανασυχούν όμω, ότι η προσπάθεια για την καταπολέμηση χρηματοδότησης των τρομοκρατιών αφορά, ε, εστιάζεται επί συγκεκριμένου στόχου και χάνουμε το γενικό στόχο. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις εδώ, σημασίας μεταξύ διαφόρων οικονομικών εγκλημάτων. Ήθελα να πω ότι συζητείτε το θέμα. Σε ποιο βαθμό μονοπολούνται οι ε, πόροι για την καταπολέμηση της χρηματοδοτής τρομοκρατών και αγνοούνται άλλοι τομείς. Και βλέπετε πώς άλλαξε ο ορισμός της μονάδας καταπολεμής οικονομικού εγκλήματος συλλογής πληροφοριών. Αρχικά θεωρούνται φορεί κατα του ξυπλήματο χρήματο. Τώρα παρουσιάζονται σαν ειδικέ μονάδε συλλογή πληροφοριών με πολλαπλά καθήκοντα. Κατά πολέμηση κοινωνική απάτη, φοροδιαφύγη, οργανωμένου κλίματο κ.ο.κ. Σημαντική αλλαγή αυτή. Σημαντική. Για το υπόλοιπο τη παρουσιάσεω να επιμένω επί τριών λειτουργιών των μονάδων αυτών. Πρώτα απ' όλα συλλογή πληροφοριών Δεύτερον, ανάλυση αυτών. Οι πληροφορίε να αναλυθούν σωστά. Και τρίτον, διάδοση πληροφοριών για τα οικονομικά. Θα αναφερθώ σε κάθε στοιχείο αυτών. Πρώτον, συλλογή πληροφοριών. Βασικό υλικό είναι εκθέσεις οικονομικών συναλλαγών που λαμβάνουν από τους φορείς υποβολής εκθέσεων και αναφορών τα χρηματοστικά ιδρύματα και κυρίως οι τράπεζες δίνουν βασικά αυτές τις πληροφορίες. Σχετίζονται επί υπόπτων συναλλαγών αυτές οι εκθέσεις. Είναι ένα μοντέλο που εδράζεται επί πονιών. Όταν υπάρχει πόνια ότι γίνεται εξέπλημα χρήματος, πρέπει αυτό να αναφερθεί στις μονάδες καταπολεμής οικονομικού εγκλήματος. Αναφέρθηκα στα χρηματοστικά ιδρύματα, μπορεί να είναι και άλλοι φορείς, όπως οι νομικοί. Όπως αναφέρεται και στη διαφάνεια, οι μονάδες καταπολεμήσεως οικονομικού εγκλήματος είναι στο σημείο επαφή οικονομικών και ασφαλείας. Οι χρηματοστικά ε, ιδρύματα δίνουν οικονομικές υπηρεσίες ε, και πληροφορίες. Δεν παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας, ούτε αστυνομικέ. Η δουλειά τους βασίζεται οικονομικά και οικονομικές συμβουλές. Αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα έχουν στόχο να αυτοπροστατευτούν από τις μυστικές αρχές και όχι από τους εγκληματίες ή τους τρομοκράτες. Θέλουν να συμμορφωθούν, να αποφύγουν κυρώσεις. Έχουν φήμη να προστατεύσουν. Θέλουν να προστατευτούν από οικονομικές κυρώσεις. τίθεται σημαντικό θέμα όσον αφορά τι πρακτικέ αναφορών. Αμυντική ενημέρωση, defensive reporting. Δηλαδή, κατατίθενται οι συναλλαγέ βάσει υπονοιών, αλλά το χρησιμοποιητικό Ίδρυμα προσπαθεί να προστατευτεί όσον αφορά τη φήμη του και τι υπόνοιε κλπ. Και να μην θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται. Αμυντικά κινούνται δηλαδή. Ίσως να υποβάλλονται υπερβολικές εκθέσεις από το φόβο υπονοιών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο Κάθε φορά που έχουν αμφιβολήσει σε χρηματοδοτικά ίδρυματα προσπαθούν να καταγγείλουν για να είναι ασφαλή. Αυτό έχει αντίκτυπο όμω όσον αφορά τον όγκο εργασία ε, των μονάδων καταπολεμήσεω εγκλήματο. Δημιουργείται περισσότερο θόρυβο και θολούρα παρά πληροφορίε να χορηγούνται. Άλλη δυνατότητα για αμυντική υποβολή εκθέσεων έχουμε υπο, υπο, λιγότερε υποβολέ όπω στην Ελβετία. Μόνο όταν υπάρχει επιλογή παρακαταγγελία όταν είναι συσυδής ο πελάτης σου, ξεσπάει σκάνδαλο όπως τα Panama Papers, κάνεις την καταγγελία σου για να μην διωχθείς μαζί με τον πελάτη σου. Αυτό αληθεύει κυρίως όσον αφορά τα φορολογικά εγκλήματα, διότι επί μακρόν τα χρηματοδοτικά ιδρύματα όλους ιδιαίτερος συμβιβαζόταν, έλεγαν θέλουμε να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα χρήματος διότι σχετίζεται με παράνομους φορείς, διακινητές, οργανωμένο έγκλημα, τρομοκράτες. Αλλά ποια ήταν η ιδέα να μην συμπεριλαμβάνουν νόμιμους φορείς ή νόμιμους οικονομικούς πολιτικούς φορείς που μπορούν να προβαίνουν σε ε, και λοιπά και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Και τίθεται θέμα εδώ, πρόβλημα, πώς να αντιμετωπίσουν αυτό. Και πώς να καταγγέλουν με αμυντικό τρόπο τα θέματα φοροδιαφυγής και φοροποφυγή. Δεύτερο στοιχείο που βλέπετε, ότι οι πρακτικές καταγγελιών μεταξύ υπονίας και οικονομικών ορίων το βασικό σύστημα που βασίζεται επί υπονοιών και θα μπορούσα να πω ότι από χώρα σε χώρα το πώς ερμηνεύεται η πόνοια ποικίλει. Εύλογη πόνοια, τεκμηριωμένη πόνοια κλπ. Και ο τρόπος που παρουσιάζεται η πόνοια καταλήγει αναλόγως σε καταγγελία και ο τρόπος ποικίλει από χώρα σε χώρα. Το βλέπει κανείς αυτό. Με τον όγκο των καταγγελιών που καταφθάνουν σε άλλες χώρες υπάρχει αυτόματη καταγγελία. Βασίζεται επί οικονομικών ορίων. Νομίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέσσερις χώρες το κάνουν αυτό. Παράδειγμα. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδάς, όλες οι ηλεκτρονικές μετα... Ε, μεταφορές χρημάτων πάνω από 10.000 δολάρια αποστέλλονται αυτόματα στις μονάδες καταπολεμής οικονομικού εγκλήματος. Άρα πέρσι στον Καναδά λάβανε 24 εκατομμύρια καταγγελίες και εκθέσεις. 100.000 βασιζόταν επί υπονοιών, οι υπόλοιπε επί αυτόματα τη κοινοποίηση των συναλλαγών. Σε ποιο βαθμό έχουμε προστιθέμενη αξία όσον αφορά την καταπολέμηση φοροδιαφυγή μέσω του αυτόματου αυτού ορίου. Παρουσιάζεται και προωθείται ότι δίνει αξία όσον αφορά την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή στον Καναδά τουλάχιστον. Διότι οι φορεί που υποβάλλουν τις εκθέσεις, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, πρέπει να υποβάλλουν τις εκθέσεις αυτομάτως από 10.000 και περισσότερες συναλλαγές άμεσα προ τι μονάδε καταπονομή του ε, οικονομικού εγκλήματο, οι φορολογικέ αρχέ ταυτόχρονα. Άρα είναι σημαντικό εργαλείο η πρόσβαση σε αυτέ τι πληροφορίε. Τώρα, δεύτερο καθήκον των μονάδων αυτών, ανάλυση πληροφοριών. Παραλάβουν πληροφορίε για ύποπτη συναλλαγή. Τι κάνουν τότε, πώ αναλύουν τι πληροφορίε πώς μεταφράζονται οι πληροφορίες σε συγκεκριμένες δράσεις και κινήσεις. Ξέρετε τη διαφορά μεταξύ των μοντέλων των μονάδων κατά καταπολεμής οικονομικού κλίματος. Έχουμε δικαστικό μοντέλο, επιβολής του νόμου, αστυνομικό μοντέλο, διοικητικό μοντέλο, διάφορα μοντέλα. Τι να πω εδώ, ότι είναι σημαντικό το θέμα του καθεστώτος, αλλά καλύπτονται και διάφορες άλλες διαφορές. Και για μονάδες που σχετίζονται με το ίδιο μοντέλο. Πρώτη μεγάλη διαφορά πρόσβαση σε εθνικές βάσεις δεδομένων και κεντρικά μητρώα. Ποικίλει κατά πολύ από μονάδα σε μονάδα, ακόμα και αν οι δύο είναι διοικητική μορφής ή επιβολή νόμου. Πάμε τώρα στην πρόσβαση στι εθνικέ βάσει δεδομένων και στα Μητρώα αργότερα, όσον αφορά τα εμπόδια, όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία. Δεύτερο θέμα, η διαφορά μεταξύ μοντέλων αναλυτικό μοντέλο και μοντέλο συλλογή των διαφόρων στοιχείων. Στην πρώτη περίπτωση, η μονάδα κατανομή του εγκλήματο μπορεί να ειδωθεί σαν βάση δεδομένων. Προσβάσιμη στου εταίρου για την επιβολή του νόμου, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν πολλοί φορεί εμπλεκόμενοι που έχουν πρόσβαση άμεση στη βάση δεδομένων των μονάδων καταπολεμή οικονομικού εγκλήματο, χωρί να γίνεται ανάλυση ειδική. Και στη ΣΥΠΑ το ίδιο γίνεται. Η αστυνομία μπορεί να ψάξει στη βάση δεδομένων άμεσα, χωρίς να υπάρξει ανάλυση πλευρά τη μονάδα καταπλωμίσεω εγκλήματο. Στον ελληνικό μοντέλο δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στον ελληνικό μοντέλο ποτέ δεν δίνεται πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Οι εταίροι επιβολή του νόμου λαμβάνουν μόνο το προϊόν τη ανάλυση. Ε, τη συλλογή των πληροφοριών από την μονάδα για το οικονομικό έγκλημα και είναι διαφορετικό. Δηλαδή τι γίνεται, δίνουμε πρόσβαση σε όλους τους εταίρους μας, αστυνομία, μονάδες πληροφοριών, φορολογικές αρχές, πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Ή υπάρχει συγκεκριμένη αποστολή που έχει μονάδα καταπολεμής του εγκλήματος να κάνει πρώτα την ανάλυση και μετά τα προϊόντα της ανάλυσης να τα διαβιβάζει. Τώρα, σχετικά με τον τρίτο βασικό, βασική λειτουργία, διάδοση πληροφοριών, να στέλνει στοιχεία προς τους εταίρους δηλαδή η μονάδα, για την καταπολέμηση συγκεκριμένων εγκλημάτων απλή ερώτηση που δεχτήκαμε. Ποιοι είναι οι πελάτε των πληροφοριών για τα οικονομικά, ποιοι είναι οι βασικοί εταίροι που παίρνουν το προϊόν στα χέρια του που συλλέγει μονάδα για τα οικονομικά. Από χώρα σε χώρα έχουμε μεγάλε διαφορέ, Φερρυπίν, Ελβετία. Μόνο οι διοκτικέ αρχέ. Άρα η μονάδα διώξεω του εγκλήματο είναι το επιχειρηματικό κλάδο τη δικαιοσύνη. Στον Καναδά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εντελώ διαφορετικά. Μπορεί να στείλουν τι πληροφορίε σε μονάδε συλλογή πληροφοριών, στην αστυνομία, φορολογικέ αρχέ κλπ, και κλπ. Και στη Γαλλία και σε κάποιο βαθμό και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν δύο μοντέλα. Δικαστικό σκοπό για δίωξη είναι ο σκοπό χρήση των στοιχείων ή για τη χρήση άλλων φορέων. Μετά, διάκριση μεταξύ ενεργού αποκαλύψεως και αντιδραστικής αποκαλύψεως. Όταν μια μονάδα λαμβάνει μια έκθεση για ύποπτη συναλλαγή πρέπει να κάνει την ανάλυση. Στέλνει άμεσα ε, αυταπάγγελτα σε εταίρο τις πληροφορίες ή περιμένει να δεχτεί αίτηση από τον εταίρο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Στον Καναδά, Φερρυπίν, πράγματι ψάχνουν στη βάση δεδομένων και βλέπουν τι ζητούν οι εταίροι. Αν οι εταίροι ζητούν συγκεκριμένο είδο αδίκημα, κάποιε πληροφορίε θα το βρουν. Δεν θα βρουν κάτι άλλο όμω. Διότι δεν κινούνται αυτεπάγγελτα. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ κρατών μέλων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Οπότε, αν κανένα εταίρο δεν ζητά κάτι για φορολογικό αδίκημα, δεν θα βρει τίποτα για το φορολογικό αδίκημα και ποτέ δεν θα στείλει κάτι. Άρα υπάρχει διάκριση μεταξύ ενεργού και αντιδραστικού όσον αφορά την προσέγγιση. Αυτεπάγγελτα και κατόπιν ετήσεως. Τώρα, όσον αφορά τη διάδοση των πληροφοριών, αλλά σε διεθνή συνεργασία. Θα το διατρέξω γρήγορα για να κλείσω όσον αφορά τα εμπόδια, μέσω των εμποδίων. Έχουμε δύο βασικέ διάβλου επικοινωνία. Πρώτα, διεθνή διάβλο όσον αφορά την ομάδα Egmont, με συγκεκριμένο διάβλο πληροφοριών. Ε, η Egmont Group είναι διεθνής οργανισμός για καταπολέμηση του εγκλήματος. 152 μονάδες συμμετέχουν εκεί στην ομάδα Egmont και έχουν το ασφαλές δίκτυο Egmont για ανταλλαγή πληροφοριών για συγκεκριμένα οικονομικά εγκλήματα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχετε το FIU-NET. Κάτι αντίστοιχο, αλλά με διαφορετικές δυνατότητες, αλλά και χαρακτηριστικά. Τώρα, γιατί θέλουν να συνεργαστούν. Μπορούν να λάβουν έκθεση για ύποπτη συναλλαγή και μπορούν να δουν ότι περιέχει κάποιο διεθνέ στοιχείο. Ζητούν από του άλλου εταίρου. Έχετε πληροφορίε γι' αυτό. Ή μπορεί να λάβουν συγκεκριμένο αίτημα από του εταίρου του σε εθνικό επίπεδο και να πούνε εντάξει, χρειαζόμαστε να παρακολουθήσουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα στο εξωτερικό. Η διαφορά μεταξύ ομάδα Egmont Group και τη FIU Nut είναι πόσο προχωρημένο είναι ο ένα και άλλο. Η Egmont Group είναι πιο προχωρημένη. Μπορεί είναι πιο εύκολο να πάει πληροφορίε άμεσα από εκεί και υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει πολυμερή συνεργασία. Όχι μόνο διμερή, πολυμερή, αλλά πολύ πιο προχωρημένη η ομάδα Egmont. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κυρίω όσον αφορά ε, το ευρωπαϊκό δίκτυο, το FIU-EU. Κλείνοντα, αν έχω χρόνο για τα εμπόδια, ποια είναι τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των μονάδων αυτών κατά περίπτωση του οικονομικού κλίματο. Πρώτα απ' όλα η έλλειψη δυνατότητα ανταπόκριση σε διεθνή αιτήματα. Ίσως δύο να πω πάνω σε αυτά, δύο πράγματα. Πρώτον, κάποιες μονάδες δεν μπορούν να λάβουν πληροφορίες άμεσα από τους φορείς καταγγελιών αν δεν έχουν συγκεκριμένη έκθεση για ύποπτη συναλλαγή στην μάση δεδομένων. Ας πούμε, η Γαλλία ζητά πληροφορίες στον Ηνωμένο Βασίλειο. Εν τη αυτή περιπτώσει, το Ηνωμένο Βασίλειο λέει δεν μπορούμε να ζητήσουμε από την τράπεζα να μα δώσει πληροφορίε, διότι δεν λάβαμε καμία υπόνοια συναλλαγή για την ίδια περίπτωση. Αυτό δεν ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μπορούσε να ισχύει για την Ελβετία. Είναι σημαντικό πρόβλημα. Αν δεν έχουν την ίδια ύποπτη συναλλαγή σε εθνικό επίπεδο, στη βάση δεδομένων δεν μπορούν να ζητήσουν για κάποια άλλη μονάδα πληροφορίε. Και η δυνατότητα να ανταποκριθεί διαφέρει ανάλογα με το έγκλημα. Μπορεί να έχει πολύ στενού εταίρου, δύο μονάδε που είναι πολύ στενέ να ανταλλάσσουν πολλά για ένα θέμα, για τα ναρκωτικά, όχι για τη φοροδιαφυγή. Οπότε το είδος του εγκλήματος και όχι το είδος των εταίρων επίσης είναι σημαντικό ζήτημα. Όσον αφορά τώρα την αυτεπάγγελτη διάδοση των πληροφοριών, την αυθόρμητη, είναι σημαντικό θέμα το οποίο τίθεται στην οδηγία, την τελευταία οδηγία. Βασικά, τι λέγεται εδώ, ότι αν μια χώρα λάβει μια έκθεση για ύποπτη συναλλαγή που σχετίζεται με άλλη χώρα, ποια είναι η ιδέα, να στείλει αυτομάτως αυτή τη χώρα πληροφορίες, αυτό δεν ισχύει για την ώρα, δεν αφορά τη χώρα μας λένε, μένει στη βάση δεδομένων, δεν δίνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει αυθόρμητη μεταβίβαση πληροφοριών προς τη χώρα που ε, σχετίζεται με τις υπηρεσίες κυρίως όσον αφορά τη φοροδιαφυγή. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Και τέλος, τελετικό στοιχείο για την καταχρηστικό περιορισμό της χρήσης οικονομικών πληροφοριών. Επιμένουμε πολύ από αυτού όσον αφορά την αδυναμία πρόσβασης στις πληροφορίες. Μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό όσον αφορά τον δι... πραγματικό δικαιούχο ιδιοκτήτη, τα μητρό όσον αφορά του κατόχου τραπεζικών λογαριασμών. Όσον αφορά την πρόσβαση, είναι ένα θέμα όσον αφορά τη χρήση οικονομικών πληροφοριών. Κάποιε χώρε, Φερρυπίν, ανταλλάσσουν πληροφορίε όσον αφορά φορολογικά εγκλήματα, αλλά θα πούν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία για θέματα φορολογικά. Αλλά λαμβάνουν τι πληροφορίε, αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για αυτό που θέλουν. Οπότε, να, για να διώξουν ή να συνεχίσουν ε, διελεύκανση υποθέσεων ξεπλήματο χρημάτων σε αποφυγή. Είναι όχι μόνο οι πληροφορίε, αλλά επί, το να επιτραπεί να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίε σε συγκεκριμένα θέματα όπω είναι η φοροδιαφυγή. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στον τελευταίο κύκλο ομιλητών που οπωσδήποτε θα ασχοληθούν με τα ζητήματα αυτά των παρουσιάσεων. Οπότε, περνάμε στους συνεισηγητές ε, τη Επιτροπής ε, Πάνα και ξεκινάμε από εσάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνολική αυτή παρουσίαση. Να ξεκινήσω με την τελευταία παρουσίαση για τις μονάδες ε, ξεπλήματος χρήματος. Θα ήθελα λοιπόν να μπορείτε να μας ε, εξηγήσετε τρία βασικά προβλήματα. Την έλλειψη πληροφοριών, το ότι άλλες μονάδες πληροφοριών έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες, άλλες μπορούν να επιβλέπουν το τραπεζικό τομέα, άλλες όχι. Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις με το ξέπλυμα χρήματος είναι ότι, ξέρετε, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν το σύστημα το χρηματοπιστωτικό για να ξεπλύνουν τα χρήματά τους και το σύστημα που έχουμε δημιουργήσει ε, είναι πολύ εύκολο τελικά για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Οπότε αν μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τα βασικά για την σύσταση μιας τέτοιας μονάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το αν θα μπορούσε να επιλύσει αυτά τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε για τις αρμοδιότητες, την αποτελεσματικότητα και τον ρόλο των μονάδων πληροφοριών. Εσείς βλέπετε μία προσέγγιση που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Έχουμε βεβαίως το δίκτυο κατά πολέμηση οικονομικού εγκλήματος, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα για να χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια ευρωπαϊκή μονάδα πληροφοριών που θα έχει και την δυνατότητα να εξετάζει το πώς οι εγκληματίες χρησιμοποιούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να εξυπλύνουν τα χρήματά τους. Δεύτερον, για την ε, συνεργασία. βέβαια, ε, ο Δανό ε, προξενεί αμηχανία το ότι οι Δανείοι δεν συνεργάζονται πλήρω ε, και θα ήθελα να σα ρωτήσω ποιο είναι ο λόγο γι' αυτό. Όχι μόνο για την Δανία, αλλά γενικώ. Και πώ λύνεται αυτό το ζήτημα με τρόπο αποτελεσματικό. Δηλαδή, εντάξει, η Επιτροπή έχει προσπαθήσει να το προσεγγίσει πολλέ φορέ, αλλά είναι νομίζω ζήτημα του ότι δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς. Και βεβαίως, γιατί η Δανία, για να πω για τη δικιά μου τη χώρα, δεν απαντάει εγκαίρως, ε, δεν απαντάει σε ερωτήσεις που κάνετε. Υπάρχει κάποιος τρόπος να βελτιωθεί η κατάσταση. Να τους ξεκαθαρίσετε ποιο είναι το, το θέμα. Σας ευχαριστώ. Έχετε... Δεν ξέρω. Θα ακούσετε την απάντηση και εσείς μπορείτε μετά να κάνετε κάποια τηλεφωνήματα στη Δανία να βοηθήσετε. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Λοιπόν, για την ε, μονάδα πληροφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν το βασικό ερώτημα. Θα έλεγα ότι υπάρχει ήδη κατά κάποιον τρόπο, η υπάρχει η δυνατότητα με το FIUNET που θα μπορούσε νομίζω να αποτελέσει μια κεντρική τέτοια μονάδα γιατί δεν ξέρω, ε, ίσως το είπα λίγο γρήγορα, αλλά με το FIUNET. Ναι, όταν ανέφερα εκεί την ιδέα της ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτό το οποίο είναι δυνατόν τώρα, σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια, είναι να κάνουμε την αυτόματη διασταύρωση. Ας πούμε, σποθέσουμε ότι μια χώρα δίνει μέρος της εθνικής βάσης δεδομένων, τη βάζει σε ένα φίλτρο και είναι διαθέσιμο στις άλλες μονάδες πληροφοριών και μπορούν αυτομάτως να τσεκάρουν. Να σας υποθέσουμε ότι η Γαλλία βάζει ένα φίλτρο, π.χ. θεματικό φίλτρο. Όλες οι αναφορές που λαμβάνουμε σε σχέση με φοροδιαφυγή τις ε, δίνουμε και έχετε όλη πρόσβαση. Εάν το κάνουν όλοι μπορούν να κάνουν κάποια διασταύρωση που δεν μπορούσαν να την είχαν σκεφτεί πριν και να ζητήσουν διεθνή συνεργασία. Ένα θέμα λοιπόν θα ήταν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες να μοιραστούν πληροφορίες ε, μεταξύ τους. Ε, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο αυτή την στιγμή και κάποιοι πραγματικά το στηρίζουν. Άλλοι δεν θέλουν γιατί το FIUNET αυτή τη στιγμή βασίζεται εντό της Europol και είναι θέμα γιατί φοβούνται την αστυνομικοποίηση της ε, μονάδας ε, πληροφοριών και για το θέμα αυτό επίσης αυτό σχετίζεται και με την εντολή της Europol. Η για την ώρα δεν ε, θεωρούν ότι πρέπει να ασχολούνται με τα φορολογικά. Ξέπλυμα χρήματος ναι, αλλά φορολογικά δικήματα όχι. Και το βλέπουμε αυτό όταν μελέτησαν τα ζητήματα του Panama Papers. Προσπάθησαν να βρουν άλλα αδικήματα, όχι φορολογικά. Και βεβαίω το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουν είναι να αναζητούν παράνομη μετανάστευση. Οπότε είναι θέμα προτεραιοτήτων, αλλά η δυνατότητα υπάρχει ήδη με το FIUNET. Μάλιστα. Ε, να είστε σύντομοι παρακαλώ. Ναι, για το θέμα της Ανίας. Κοιτάξτε, τέλος Μαρτίου ζητήσαμε τη συνεισφορά που έλπε και η Δανία, η Κροατία και η Ισπανία υποσχέθηκαν να μου απαντήσουν μέχρι τα μέσα Απριλίου. Αναμένουμε. Ε, έχουμε αργήσει λίγο, αλλά αν μπορείτε να μας βοηθήσετε θα το εκτιμούσαμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία. Περνάμε λοιπόν ε, στον άλλο συνεισηγητή, τον κύριο Πίτερ Γεζεκ και να σας υπενθυμίσω ότι όσο συντομότερη ερώτηση τόσο περισσότερο χρόνο έχουμε για να απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Ακόμα... Θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Ο συνάδελφος που έφυγε υπενόησε ότι υπάρχει ένα άκαμπτο συγκεντρωτικό σύστημα, αλλά αυτά τα οποία ακούμε ε, δείχνουν μια ξεκαθαρά διαφορετική εικόνα. Αντιθέτως φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ χαλαρή, με μεγάλη ευελιξία για τα μέλη της τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα, γιατί αυτό το οποίο ακούσαμε για τις ε, συνεισφορές των κρατών μελών ε, στην μελέτη ήταν πολύ ενισχυτικό και δυστυχώς επιβεβαιώνει το χαμηλό επίπεδο συνεργασίας με τα κράτη-μέλη, την έλλειψη βούλησης για να δώσουν δεδομένα όταν τους ζητούνται και επιπλέον επιβεβαιώνεται ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις στα κράτη-μέλη για το πώς θα αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά. Οπότε Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση στις ε, συστάσεις μας. Μια συγκεκριμένη ερώτηση για τις μονάδες πληροφοριών και την συνεργασία τους με τις φορολογικές αρχές μας. Είπατε ότι δεν είναι ιδανική. Η συνεργασία μεταξύ FAU και των ε, μονάδων πληροφοριών δηλαδή και των φορολογικών αρχών και άλλων αρχών. Ε, τι μπορεί να γίνει δηλαδή και υπάρχει κάποια χώρα που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα υπόδειγμα ας πούμε. Ευχαριστώ. Ωραία. Τρία λεπτά έχετε για να απαντήσετε. Ναι. Θα ήθελα να απαντήσω την ερώτηση για τις μονάδες πληροφοριών και τις φορολογικές αρχές γιατί ήταν στην αρχική ανάλυση της έκθεσης. Στην έκθεση περιγράφουμε διάφορους τρόπους συνεργασίας μεταξύ μονάδων πληροφοριών και φορολογικών αρχών. Ένα θέμα είναι αυτό το οποίο αναφέρουμε, οι πολλαπλές εκθέσεις. Αυτό το οποίο περιέγραψε μόλις ο Αντωνίου, ότι δηλαδή οι εκθέσεις υπόπτων συναλλαγών δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από μονάδε πληροφοριών αλλά και από άλλε αρχέ και υπάρχει έτσι ένα πρόβλημα όταν δύο αρχές ερευνούν το ίδιο συμβάν. Και στην έκθεση εμείς χρησιμοποιούμε μια άλλη έκθεση του ΩΣΑ που αναλύει το διαφορετικό επίπεδο συνεργασίας μονάδων πληροφοριών και φορολογικών αρχών και μας δίνει ενδιαφέρουσες ιδέες. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής συνεννόηση, ένα μνημόνιο μεταξύ των αρχών ή να υπάρχουν σύνδεσμοι της μίας αρχής στην άλλη και βεβαίως να προωθούμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και κάποιο είδου κατάρτιση. Οπότε υπάρχουν τρόποι να βελτιώσουμε την λειτουργία και υπάρχει και είναι και μέσα στην έκθεση. Δεν ξέρω, Αντώνιο, αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Ε, ναι, είπε είναι σαφώς κάτι το σημαντικό. Ε, πάντα μας λένε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή λένε πριν είχαμε το λεγόμενο συνικό τείχος, τώρα έχουμε απλά το τείχος του Βερολίνου. και βεβαίως αυτό σχετίζεται και με την ιστορία της καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος γιατί σχετίζεται με την παράνομη διακίνηση, το οργανωμένο έγκλημα και βεβαίως ε, υπάρχει ακόμα αυτή η νοοτροπία όσον αφορά τις μονάδες πληροφοριών που διαφέρει βεβαίως από τις φορολογικές αρχές. Και είναι δύσκολο για τις φορολογικές αρχές να συνεργαστούν με εισαγγελείς ε, γιατί θεωρούν ότι το βασικό ζήτημα είναι διοικητικό Οπότε υπάρχει και ζήτημα ε, νοοτροπίας διαφορετικής, ακόμα και αν είναι εκείνη η αρμοδιότητα. Ευχαριστώ. Ο Ντάριο Ροζάτη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να εκφράσω τις ε, ευχαριστίες μου στους ομιλητές ε, για τις προσπάθειές τους και τα συμπεράσματά τους. Η πρώτη μου αντίδραση σε αυτά τα οποία είπατε είναι ότι δεν υπάρχει αναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών. Τα μοντέλα, οι διαδικασίες, το πεδίο η θέληση συνεργασίας και βεβαίω αυτή η ποικιλομορφία εκτείνεται και στην συνεργασία μεταξύ αυτών και των φορολογικών αρχών. Η πρώτη ερώτηση είναι σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει την οδηγία της εφαρμογής για το ξέπλυμα χρήματος, τις οδηγίες. Πώς μπορεί δηλαδή να φροντίσει τα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη εκπληρώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις ύποπτες συναλλαγές, πώς μπορούν να γίνουν αντιληπτές αυτές οι ροές όταν το νομικό και διοικητικό πλαίσιο είναι τόσο διαφορετικό. Και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι εφαρμόζεται σωστά η οδηγία ξεπλήματος χρήματος τρόπο που εγγυάται την εκπλήρωση των στόχων της. Και το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Όταν έχουμε το μοσαϊκό ε, νομοθεσίας ε, υπάρχει ο πειρασμός να σκεφτούμε ότι σε κάποιες χώρες είναι απλά ευκολότερο να φοροδιαφύγει κανείς. Και αυτό επιβεβαιώνεται νομίζω και από τα στατιστικά στοιχεία των Panama Papers, γιατί κάποιες χώρες εμφανίζονται εκεί πιο συχνά από άλλες. Αν ισχύει αυτό, τότε η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και το προηγούμενο πάνελ ότι κάνουμε προβολή ας πούμε, από την αναλογία των παράνομων συναλλαγών ε, ή την ε, υστέρηση των φορολογικών εσόδων σε σχέση με τα συνολικά φορολογικά έσοδα και από αυτό αυτή την αναλογία την προβάλλουμε σε άλλες χώρες ε, δεν έχει πολύ νόημα έτσι γιατί αν υπάρχουν αυτές οι διαφορές, οι θεσμικές, εξορισμού, ε, θα είναι διαφορετική και η αναλογία στέρησης φορολογικών εσόδων σε κάθε χώρα. Μπορείτε να πείτε κάτι από αυτό. Για την πρώτη σας ερώτηση, για την έλλειψη αναρμόνησης και μετά πώς να παληθεύσουμε κατά πώς εφαρμόζεται αφορμόζεται η οχι και αν εφαρμόζεται και αποτελεσματικά. Είναι και αυτό ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχει συμμόρφωση. Οι μονάδες δηλαδή αυτές οικονομικών πληροφοριών κάνουν τη δουλειά τους. Έπειτα υπάρχει και το θέμα της τεχνικής συμμόρφωσης. Έχετε πληροφορίες, τις αναλύετε, φροντίζετε να τις διαδώσετε. Δεύτερον, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Ε, είναι όλο το θέμα καταπολέμησης της νομοποίησης παράνομου χρήματος. Τι σημαίνει να εφαρμόσετε αποτελεσματικά η οδηγία. Θα πάρετε διαφορετικές απαντήσεις. Για το Ηνωμένο Βασίλειο θα σας πει εμείς έχουμε 400.000 αναφορές για υπόνοιες, ενώ μια άλλη χώρα θα σου πει εμείς έχουμε μόνο 2.000. Οπότε, τι θα απαντήσουν αυτοί που παίρνουν μόνο τις 2.000 θα πούνε ότι είναι αποτελεσματικοί γιατί έχουν προχωρήσει στην επεξεργασία 80%. Και είναι χρήσιμο. Φτάνει στον τύπο υπόθεση. Αν έχει φτάσει στον τύπο υπόθεση, προφανώς και οι μονάδες αυτές θα αντιδράσουν. Το βασικό όμως είναι να δούμε ποια είναι τα κριτήρια για να εντοπίσει κανείς την αποτελεσματικότητα. Κάποιος θα πει έχει να κάνει με τον αριθμό διώξεων. Όχι, άλλος θα πει έχει να κάνει με τις πληροφορίες και θα πούνε εμείς είμαστε ε, μονάδα πληροφοριών. Άρα πρέπει αλλιώ να μας αξιολογήσετε, όχι από τον αριθμό των διώξεων, αλλά από τον αριθμό των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει. Άρα λοιπόν πρέπει κανείς να προσπαθήσει να καταλάβει το έργο τους, γιατί είπαμε ότι πάμε από τη φοροδιαφυγή μέχρι τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας δεν λέω ότι είναι άσχετη ερώτηση, απλώς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Η άλλη ερώτηση που είχε να κάνει με τη μεθοδολογία. Κοιτάξτε. Στην μελέτη μας θα κοιτάξουμε τι γίνεται σε όλες τις χώρες μέλη. Αλλά όπως είπε ο συνάδελφος, θα είναι περιορισμένο. Κοιτάμε τα νούμερα του προσωπικού που δουλεύει σε αυτές τις μονάδες οικονομικών πληροφοριών, τον αριθμό των υποθέσεων που επεξεργάζονται, τις περιπτώσεις όπου έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Είναι περίπλογο να πούμε ότι αυτή η χώρα είναι αποτελεσματική. Αυτή η χώρα δεν είναι αποτελεσματική. Αλλά θα συγκρίνουμε όλε τις χώρες μέλη. Ο κ. συγγνώμη, η ερώτησή μου ήταν κάπως διαφορετική. Εκτιμήσατε τις απώλειες από τα φορολογικά έσοδα στις διάφορες χώρες. Είπατε ότι δεν έδωσαν στοιχεία όλες οι χώρες και άρα πήρατε στοιχεία από μερικές μόνο χώρες και αυτές τις προβάλλατε και στις υπόλοιπες. Κάνοντα την υπόθεση ότι υπήρξε ίδια απώλεια εσόδων παντού. Εφόσον όμως είναι τόσο διαφορετικά τα συστήματα και τόσο περίπλοκη η κατάσταση, εγώ νομίζω ότι η υπόθεση αυτή, ότι το ίδιο ισχύει και στι υπόλοιπε, οπότε προβάλλατε τα στοιχεία και στις υπόλοιπε, δεν ε, στέκει. Πρόεδρο, δεν είναι βέβαια αυτό που εξετάσατε εσεί αυτό το πάνελ. Ίσως θα έπρεπε αυτό να το συζητήσουμε με του προηγούμενου ερευνητέ. Τώρα, ο κύριος Ρωμόνατον από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Ισπανία. Ισπανικά. Οπότε βάλτε τα ακουστικά σας. Λοιπόν, θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτά που μας είπατε και έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι, δηλαδή, όπως ο κύριος Ρωσάτη και εκπρόσωπος της Άλντε, είπαν ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές από αυτά που μας είπατε εσείς δηλαδή μεταξύ των χωρών μας. Υπάρχουν ε, βέβαια πολλές διευκολύνσεις για να γίνονται ανταλλαγές πληροφοριών, αλλά η αίσθηση που έχω είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που μας λείπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μία μονάδα παρακολούθησης, ελέγχου, ενημέρωσης για όλες τις εθνικές φορολογικές πολιτικές. Η ερώτηση ίσως δεν είναι για σας, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει να το γνωρίζουμε, γιατί θα μπορούσε να είναι σύσταση της Επιτροπής μας. Μήπως πρέπει να ζητήσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μια τέτοια μονάδα ελέγχου και παρακολούθησης ε, των πληροφοριών, ώστε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και να φροντίσουμε έτσι να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα της διαφοράς στην νομοθεσία μας. Τώρα όταν αυτές οι μονάδες οικονομικής, ε, οικονομικών πληροφοριών φτάνουν σε ένα φορολογικό παράδεισο ή σε μια δίκηση σκοτεινή η οποία δεν θέλει να συνεργαστεί και δεν ενημερώνει, τι φοβάται. Φοβάται πιο πολύ αυτές τις μονάδες οικονομικών πληροφοριών ή τελικά το παραδοσιακό δικαστικό σύστημα. Όταν αυτές οι μονάδες έχουν μια απάντηση πιο συνεργατική τι γίνεται. Και τρίτον, από την εμπειρία που έχετε εσείς στην παρακολούθηση του φορολογικού εγκλήματος, στο 80% του χρήματος που διακινείται μέσω των φορολογικών παραδείσεων έχει να κάνει με το έγκλημα και μόνο το 20% προέρχεται από φορολογική, από φοροδιαφυγή. Είναι σωστό αυτό που λέω, στέκει. Ευχαριστούμε για να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για τα σχόλια και την ερώτησή σας. Όσον αφορά τη συνεργασία των ε, μονάδων οικονομικών προφοριών ε, με εθνικές δικήσεις που δεν συνεργάζονται. Εδώ υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Όσον αφορά τα Panama Papers, η δυσκολία είναι να εντοπίσει κανείς τον δικαιούχο ιδιοκτήτη. Γιατί τελικά λέμε ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε ε, με την ε, ροή αυτή και να την ταιριάξουμε με ένα όνομα, με μια οντότητα. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Ενώ στον ε, Καναδά έχουν μεγάλες δυσκολίες να εντοπίσουν τις καναδικές εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε άλλους από το εξωτερικό. Και το άλλο ζήτημα σχετικό με τη δικαιοδοσία αυτή είναι πώς χρησιμοποιείται η πληροφορία. Υπάρχει η πληροφορία, αλλά μερικές φορές δεν έρχεται έγκαιρα ή δεν μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιήσει για φορολογικά. Υπάρχει πληροφορία, αλλά δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. Δεύτερον, για τα νούμερα. Το 80% που συνδέεται με το έγκλημα και το 20% με τη φοροδιαφυγή. Δεν το έχω ε, μελετήσει αυτό, αλλά υπάρχει το έργο του Γκαμπριέλ Τζούκμαν όσον αφορά την φοροδιαφυγή με μια νέα ε, μεθοδολογία και καταλήγει σε αυτό. Το, το 80% είναι παράνομο χρήμα και το 20% όχι. Το μικρόφωνο σας κλείστε, κύριε Τόν. Ωραία. Α, συγγνώμη, έχω μια ερώτηση ακόμα, γιατί θέλω να πω στις κυρίες που μας ενημέρωσαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι εγώ έχω πει στην Ισπανική κυβέρνηση ότι κακώς δεν στέλνει τις πληροφορίες της ε, στην ε, στις υπηρεσίες σας. Τους το έχω επισημάνει. σε ευχαριστούμε πολύ που το κάνατε. Τώρα, παρακαλώ εσείς. Το θα μιλήσω γερμανικά. Η πρώτη μου ερώτηση απευθύνεται στην κυρία Σέρε. Εάν κατάλαβα καλά, είπατε στις εισαγωγικέ σας παρατηρήσεις πως κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων είδατε ποιες δυνατότητες έχουν τα κράτη-μέλη να ανταλλάξουν πληροφορίες. Είτε δεν το είπατε μετά στην παρουσίαση, είτε μου διέφυγε. Λοιπόν, εάν δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποστείλουν επιπρόσθετες πληροφορίες, θα ήθελα να μάθω εάν τα κράτη-μέλη ε, βλέπουν κάποιες εξελίξεις, ε, π.χ. μια βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ φορολογικών αρχών και μονάδων πληροφοριών ή και της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ μονάδων πληροφοριών. Υπάρχει, υπάρχει αυτό το οποίο είπατε ότι με έθιξε κάπως και ως Γερμανό ότι πριν υπήρχε το συνικό τείχος και μετά το τείχος του Βερολίνου. Εγώ ως Γερμανός δεν ξέρω, νομίζω ότι πιο εύκολα μπορούσε να περάσει κανείς το συνικό τείχος παρά το τείχος του Βερολίνου. Λοιπόν, θα ήταν σημαντικές αυτές οι πληροφορίες για εμάς. Πού βλέπετε πρόοδο και πού βλέπετε στασιμότητα ή και νέα εμπόδια. Επιπλέον, νομίζω ήδη παρουσιάστηκε το ότι βλέπετε κάποια μοτίβα θα έλεγα ή κάποιους συσχετισμούς αλλά νομίζω ότι σημαντικό θα ήταν να ρωτήσουμε τις αρχές των κρατών μελών ποιες ήταν κατά τη δικιά τους εκτίμηση τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία οπωσδήποτε δεν θα μπορέσουμε να τα λύσουμε όλα αλλά θα έχουμε τουλάχιστον μια ιεραρχία των προβλημάτων για να επικεντρωθούμε στα σημαντικότερα και εκεί έχουμε εντύπωση πως ένας υποψήφιος, ένα υποψήφιο μεγάλο πρόβλημα ε, είναι πιθανώς ε, η στελέχωση των ε, μονάδων πληροφοριών και πιθανώς των φορολογικών αρχών. Δηλαδή είναι τεράστιοι αριθμοί ύποπτων συναλλαγών που κανείς δεν μπορεί λογικά να επεξεργαστεί. Οπότε αφενός το θέμα είναι αν η στελέχωση και οι πόροι επαρκούν και δεύτερον υπάρχουν πιθανώς διαδικασίες έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια διαλογή των πληροφοριών. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα με ενδιέφερε το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι το εξής ε, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε έναν πρωτόγονο δίκτυ, π.χ. ένα όριο των 10.000 ευρώ ή και κάποια μοτίβα σε συναλλαγές, π.χ. ποιος ε, είναι ο παραλήπτης ή ποια είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, για να μπορούμε να ψάχνουμε ας πούμε, με τρόπο με, απλό μέσω υπολογιστών και να βγαίνουν τα πράγματα. Νομίζω ότι ε, με τέτοια φίλτρα στις ε, πληροφορίες θα μπορούσαμε να ανοιχνεύσουμε περισσότερες ύποπτες συναλλαγές. Τέλος, ένα ερώτημα. Κύριε Λούκε, ε, θα, θα έχουν μετά ένα λεπτό μόνο για απάντηση έτσι που τα πάτε. Καλώς, τότε σταματάω. Λοιπόν, για να επανέλθω σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη θα δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Αυτό βάσει το ερωτηματολογίου, όχι μέσω των ε, μονάδων οικονομικών πληροφοριών. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που θα κάνουμε θα είναι όταν θα είναι έτοιμο το δελτίο της χώρας, κατά χώρα όταν έχουν ολοκληρωθεί, θα τα διαβιβάσουμε στα κράτη-μέλη, ώστε να σχολιάσουν, να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες και το ότι όλες οι απαντήσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα πάνω είναι κάτι που βοηθά τα κράτη-μέλη να δουν τι πληροφορίες δίνουν τα άλλα κράτη-μέλη και έτσι αυτό δίνει ένα κίνητρο να ιτεθούν οι καλύτερες δυνατές πληροφορίες. Κάτι για τις μονάδες οικονομικών πληροφοριών. Ε, τον Ιανουάριο έδωσε ένα έγγραφο σχετικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φωτογραφίζει το πώς ε, οι μονάδες οικονομικών πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ενετόπισαν τα εμπόδια. Έγινε η χαρτογράφηση λοιπόν βάσει ερευνών που αποστάλησαν σε προσωπικό των μονάδων οικονομικών πληροφοριών. Οι απαντήσεις δίνουν μια καλή εικόνα το πώς αισθάνονται οι μονάδες αυτές όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ τους. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς λόγω χρονικών περιορισμών δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Α, η ομάδα Άλντε δεν ζήτησε να μιλήσει εκτός τον Πίτερ Γιάζεκ. Υπάρχει κάποιος από την Άλντε που θέλει να πάρει το λόγο. Καλώς. Επόμενος. Γκουε, NGL, NGL. Εγώ. Μα χρησιμοποιήσετε εσείς το σφυράκι αν ξεπεράσει το χρόνο μου. Πρώτη ερώτηση. Δόκτωρ Μισελ, είπατε στη μελέτη ότι η Ελβετία, π.χ., δεν έχει εκθέσεις για ύποπτε συναλλαγές, δεν μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικέ πληροφορίε. Στον αναγνωστήριο είδαμε και για προφανεί λόγου, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειε, είδαμε ότι υπήρχαν κάποιε κατηγορίε επαγγελμάτων, νομικών ε, επαγγελμάτων, που είχαν πολύ χαμηλό αριθμό καταγγελιών στα κράτη-μέλη όσον αφορά τις ύποπτες συναλλαγές. Είδατε να υπάρχει κάποια μεροληψία, είδατε κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα να μην αποδίδει καλά όσον αφορά την ποσότητα καταγγελιών για ύποπτες συναλλαγές. Πώς αυτό επηρέασε τη μελέτη σας. Ε, δεύτερον, είχα μια απλούστατη ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσοι λογαριασμοί στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα είχαν παγώσει λόγω ύποπτων συναλλαγών. Συναλλαγών που σχετιζόταν με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Είχαμε δήλωση βρετανική τράπεζα τη HSBC που είχαν αρκετές τέτοιες ε, αναφορές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου είπε ότι δεν είμαστε μονάδα επιβολής του νόμου, θα πρέπει να ζητήσετε από τις ε, μονάδες οικονομικών πληροφοριών. Πήγαμε λοιπόν στον Ηνωμένο Βασίλειο και ζητήσαμε από το Βρετανικό FIU να μας δώσουν πληροφορίες. Αυτοί μας είπαν αυτό δεν είναι στην εντολή μας, αφορά κάποιο Υπουργείο, δεν θυμάμαι ποιο ακριβώ Είδατε τέτοιο πρόβλημα αρμοδιοτήτων και αυτό τι ρόλο παίζει σε αποτελεσματική ανταπόκριση όσον αφορά τα προβλήματα και στον τομέα της χρηματοδοτήσεως ε, της τρομοκρατίας. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση και τις ε, νομικές διατάξεις, επί μακρόν η συμπερίληψη α, των επαγγελμάτων, των νομικών επαγγελμάτων ήταν ε, στον τομέα αυτό. Τι είδαμε όσον αφορά τις πρακτικές τους, όσον αφορά τις καταγγελίες είναι χαμηλό το ποσοστό καταγγελιών και είναι αμυντικές καταγγελίες. Εν τη ενή υποβολή ελαχίστων ε, εκθέσεων. Περισσότερες φορές καταγγέλουν όταν δεν έχουν επιλογή, όταν ο πελάτης τους καλύπτεται από τα ΜΜΕ ή τους καλεί αστυνομία ζητώντα πληροφορίες στον πελάτη. Ξέρουν τότε ότι ο πελάτης θα διωχθεί πιθανότατα, οπότε στέλνουν αναφορά. Άρα προσπαθούν να αυτοπροστατευτούν. Δεν προσπαθούν να συνεισφέρουν στο σύστημα. Εξακολουθούν να θεωρούν ότι δεν είναι νόμιμα σωστό να συμπεριλαμβάνονται αυτοί στον μηχανισμό ξεπλήματος, κατανοήσεις του ξεπλήματος του χρήματος. Τώρα, πόσοι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν παγώσει για χρηματοδότηση τρομοκρατών. Έχετε δίκιο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη. Ε, για να έχουμε κατάλογο ονομάτων πόσοι άνθρωποι θεωρούνται ως ύποπτοι αλλά όχι πόσοι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν ε, παγώσει. Δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Να πω ε, στα γρήγορα ότι είναι σημαντικό θέμα αυτό και για τις τράπεζες το να εντοπίσουν και να μπλοκάρουν λογαριασμούς διότι είναι σημαντικό πρόβλημα να πούνε, να βρούνε ότι κάποιος είναι στη μαύρη λίστα, ότι είναι κακός και πρέπει να παγώσουμε το λογαριασμό του. Έχουν δυσκολίες εντοπισμού και ταυτοποίησης τράπεζας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος. Η κυρία Ζουλή για τους πρασίνους, αν απουσιάζει, ο υποψιάζομαι ότι θα μιλήσει. Ευχαριστώ. Η Εύα έπρεπε να φύγει. Να πάρει το τρένο για το Παρίσι. Οπότε εγώ μιλάω. Ευχαριστώ πολύ. Ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο οι απαντήσεις που δεν δόθηκαν από τα κράτη-μέλη τι θα κάνετε, θα τους στείλετε και άλλες ερωτήσεις. Αυτό είναι μέρος του εγχειρήματο ή δεν είπα το κάνουμε εμείς. Ούτω ώστε να μας δώσετε σαφή ένδειξη τι δεν έχει απαντηθεί, αυτό θα θέλαμε. Και τι έχει απαντηθεί. Ούτω ώστε να τους κυνηγήσουμε με επιστολές Μπορείτε να μου εξηγήσετε ποια είναι η διαδικασία. Δεύτερον, όσον αφορά το θέμα το άλλο, ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ μονάδων οικονομικών πληροφοριών. Θεωρείτε ότι πει, ξεπέρασαν οι μονάδες αυτές, αυτό προβλέπεται νομικά, αρνούμενες συνεργασία. Θεωρείτε ότι παραβιάζεται η νομοθεσία ή κακή διαχείριση. Τέλος, με ενδιέφερε πολύ αυτό που εξηγούσατε περί διαφορετικών ορισμών. Κατά πόσο φορολογική απάτη είναι ποινικό αδίκημα, αν είναι ένα αδίκημα που προηγείται του ξεπλήματος χρήματος. Και είδαμε ότι υπάρχει ένα όριο όσον αφορά την νομική συνεργασία, όσον αφορά το μέγεθος της φορολογικής απάτης. Μπορείτε να μας δώσετε στοιχεία Ποιος είναι ο ορισμός. Πότε η φορολογική απάτη θεωρείται σαν ποινικό αδίκημα στα κράτη-μέλη. Ποιο είναι τα όρια. Το Λουξεμβούργο έχει 200.000 ευρώ και με δυσκολία μπορείς να αποδείξεις περισσότερες περιπτώσεις ότι έχει διαπραχθεί τέτοιου μεγέθους απάτη. Άρα δεν δίνει νομική αρρωγή του Λουξεμβούργου. Από την πλευρά ξεπλήματο χρήματο, όσον αφορά υπόπτε συναλλαγέ και υποβολή εκθέσεων από αυτού και καταγγελίε αυτών. Είναι λογικό όταν δημιουργηθούν υπεράκτιες ε, εταιρείε ότι αυτές δεν ε, δημιουργούν υπόνοιες, ότι αυτή η πράξη δημιουργεί υπόνοιες, οπότε θα έπρεπε να χρησιμοποιείται σαν γενοσυργός αιτία για ε, καταγγελία περί ύποπτης συναλλαγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα για την πιθανή παράνομη συναλλαγή σε μία μονάδα πληροφοριών. Εδώ πέρα είναι νομικό ζήτημα, γιατί θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να ανταλλάσσουν πληροφορίε. Σε διεθνέ επίπεδο δεν πρέπει, μπορούν. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί είναι πληροφορίε. Δεν είναι κάποια συμφωνία στο επίπεδο της δικαιοσύνης, οπότε δεν μπορεί να είναι παράνομο, γιατί έχουν τη δυνατότητα να πούν ναι ή όχι ε, στο διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν βεβαίως κάποιες ε, καταχρήσεις που είδαμε στη διάρκεια της ε, παρουσίαση και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη. Ε, βασικά υπάρχει εξαίρεση ότι μπορεί κανείς να πει ότι είναι ευαίσθητες πληροφορίες, θέλουμε να προστατεύσουμε πολιτικούς αντιπάλους και μετά είδαμε ότι χρησιμοποιούν πολύ αυτές τις εξαιρέσεις για να αποφύγουν την συνεργασία και προφανώς γίνεται κατάχρηση. Αλλά τις περισσότερες φορές μπορούν να απαντήσουν και απαντάνε και λένε άγνωστος ή λένε ε, γνωστός και τελεία. Όσον αφορά τα οχήματα ειδικού σκοπού και τις υπερακριστηρίες, κοιτάξτε υπάρχει μία διάκριση στον νόμο μεταξύ ε, κινδύνου και υποψίας. Π.χ. οι εταιρείε offshore είναι υψηλού ρίσκου, που σημαίνει ότι θα παρακολουθούνται θα ελέγχονται περισσότερο κτλ. από τις τράπεζες π.χ. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ύποπτες ε, αυτομάτως. Ε, σχετίζονται με τον κίνδυνο, αλλά όχι ε, κάτι το οποίο γύρει υποψίες αυτομάτως. Απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις. για να απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση για την συνέχεια που θα δοθεί. Όταν λοιπόν βλέπε, θα βλέπει κανείς το δελτίο στην οθόνη και θα είναι έτοιμο, το στέλνουμε στα κράτη-μέλη, να δούμε αν θέλουν να προσθέσουν πληροφορίες. Και βέβαια αν θέλουν να κάνουν περισσότερες ερωτήσεις, ευχαριστώ και η γραμματεία επίσης ε, υπενθυμίζει συνεχώς ότι πρέπει να λάβουμε τα δεδομένα. Νομίζω ότι θα είστε και στην διάθεσή μας για περαιτέρω ερωτήσεις. Ε? Ο επόμενος είναι ο κύριος David Corbin για το EFTD. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι απαραίτητη η καταπολέμηση της εγκληματικότητας και αναγκαία. Αλλά αν μιλάμε για το κράτος δικαίου, πρέπει και η ιδιωτική ζωή και το τεκμήριο αθωότητας να γίνονται σεβαστά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κανείς αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Στα βοναπαρτικά κρατή πρέπει κανείς να αποδείξει την αθωότητά του. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη ε, βρετανικού επίπεδου. Φοβάμαι λοιπόν πως ε, ειδικά η έλλειψη ιδιωτικότητα θα οδηγήσει σε αποτελέσματα τα οποία δεν επιθυμούμε, όπως η χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη ή μετακόμιση ατόμων και επιχειρήσεων σε φιλικότερα ρυθμιστικά καθιστώτα. Όμως μπορούμε να καταπολεμήσουμε ε, την γκρίζα και τη μαύρη οικονομία με το να κάνουμε τα καθιστώτα μας φιλικότερα. Εάν επιβάλλουμε φόρο μερισμάτων και ΦΠΑ που είναι μίνιμουμ 15% ε, λογικό είναι να θεωρούν οι επιχειρήσει ότι δεν αγοράζουν τίποτα με τα λεφτά και τους φόρους που πληρώνουν. Θεωρείτε ότι ε, το να χαμηλώνουμε τους φόρους είναι πιο υποφελές για την κοινωνία από το να εφευρίσκουμε όλο και πιο περίπλοκους τρόπους εκθέσεων. Ε, χρησιμοποιούμε συνεχώς την τρομοκρατία, αλλά έχουμε φτάσει σε έναν κόσμο οργουελικό και είναι μια πολύ καλή δικαιολογία αυτή για να χώνεστε εκεί που δεν σας παίρνουν. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Το θέμα της ιδιωτικότητας είναι μεγάλο θέμα όσον αφορά το ξέπλυμα του χρήματος γιατί ήταν το, το επιχείρημα ευθύς εξ αρχής, ότι δηλαδή ε, η ιδιωτικότητα ήταν ταυτόσιμη με το τραπεζικό απόρριτο. Ε, και κάποιες χώρες δεν ήθελαν να αναλάβουν μέρος γιατί ήταν παραβίαση του τραπεζικού απορρίτου. Με την ε, Διεθνή Σύσταση του 1991 υπήρξε μια μετακίνηση μακριά από αυτό, ότι ναι βεβαίως υπάρχει τραπεζικό απόρριτο, αλλά με κάποια όρια αναφοράς με βάση κάποιες υποψίες. Αντιλαμβάνουμε ότι είναι ακόμα ένα ζήτημα σημαντικό αλλά οπωσδήποτε σχετίζεται με την εφαρμογή του ξεπλήματος χρήματος. Υπήρχε δηλαδή μια απόφαση που λέγανε ότι υπάρχει ε, τραπεζικό πόρτο μέχρι τη στιγμή που υπάρχει υποψία για ξέπλυμα χρήματος κτλ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα ζήτημα πράγματι γιατί σχετίζεται με την ε, σχέση που πρέπει να υπάρχει ε, μεταξύ παρακολούθησης ε, και ιδιωτικότητας. Απάντηση. Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι μεγάλο κομμάτι της δημοκρατίας να μπορεί κανείς να απολαμβάνει τα λεφτά του τα οποία έβγαλε εργαζόμενο σκληρά και βεβαίως είναι εύκολο για τους γραφειοκράτες ε, ειδικά στι ευρωπαϊκέ δικαιοδοσίες να ζητάνε από κάποιον να αποδείξει ότι είναι αθώος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάποιο αθώος μέχρι να αποδειχθεί ένοχο. Οπότε ε, στα δικά μα τα μάτια το σύστημά σα είναι τελείω αντιδημοκρατικό και το να δεσμεύετε τα λεφτά του κόσμου. Δηλαδή αν υπάρξει διαρροή κεφαλαίων ε, αξίζει για να προστατευτεί η ελευθερία του ατόμου. Και γι' αυτό άλλωστε φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλετε να απαντήσετε ένα μικρό σχόλιο γιατί υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ το ένα αφορά τις μαύρες λίστες ε, και το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων το άλλο θέμα που αναφέρατε είναι η ιδιωτικότητα και βασικά ως προς αυτό επανερχόμαστε στην αρχή της συζήτησης και νομίζω ε, την Επιτροπή για τα έγγραφα του Παναμά γιατί το βασικό ζήτημα ήταν μπορούμε να ακολουθήσουμε τα λεφτά, αλλά να μην τα ταυτίσουμε με συγκεκριμένη ταυτότητα και όνομα. Και αν επανέλθουμε στο θέμα του τραπεζικού απορρίτου, ε, κατά βάση δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Ε, ε, οδηγούμαστε σε μια ταυτολογία δηλαδή. Αν δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε την πληροφορία με τα άτομα, δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε το ε, Κοιτάξτε, ε, αν είναι να κάνουμε λάθος, σας είναι υπέρ της ελευθερίας. Λοιπόν, ε, θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να υπερασπιστούμε και τα συμφέροντα των σκληρά εργαζομένων που πληρώνουν φόρους και να κυνηγήσουμε αυτούς που δεν πληρώνουν. Και τα Panama Papers νομίζω έδειξαν διάφορους τρόπους ε, σκληρά εργαζομένων όπως ε, κυκλώματα πορνείας, παιδικής πορνείας κτλ. Οπότε, ο επόμενος ομιλητής θα είναι από ένα βοναπαρτικό καθεστώς. Α, δεν είναι εδώ όμως από το ΙΕΝΕΦ Οπότε, προτείνω να περάσουμε στο ΕΛΚ. Δεν. Ε, μας έχουν πει ποιος θέλει το λόγο. Οπότε, περνάμε, μπορούμε άρα να ολοκληρώσουμε. Πριν ολοκληρώσουμε, προτείνω να δώσουμε τον λόγο στους συνεισηγητές για κάποιες ε, τελευταίες παρατηρήσεις, αν το επιθυμούν. Για ε ε, έχετε τίποτα να προσθέσετε. Πολύ σύντομα. το ενδιαφέρον κομμάτι είναι να παρακολουθήσουμε τι γίνεται στις χώρες μέλη και αυτό θα γίνει με συνεργασία. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την έλλειψη συνεργασίας. Ίσως πρέπει να το βάλουμε στην έκθεσή μας. Και το θέμα των μονάδων οικονομικών πληροφοριών, όντως, πολύ τροφή για σκέψη μας δώσατε. Σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε αυτά που μας είπατε στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Φάμπιο. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέρφους εδώ για τις παρουσιάσεις τους. Ήδη έχω κάνει κάποιες γενικές παρατηρήσεις για την κατάσταση στις χώρες μέλη. Και άλλοι συνάδελφοι το έκαναν. Θα δώσουμε σίγουρα ιδιαίτερη προσοχή στα όσα μας είπατε και στις συστάσεις σας όταν θα συντάξουμε την εκθεσή μας. Πρόεδρος, Ωραία. Φτάνουμε στο τέλος. Να πιστήσω την προσοχή σας ότι 2 Μαΐου την επόμενη εβδομάδα στις 3 θα συνεδριάσουμε και πάλι με τρεις νέες μελέτες για τροφή, για σκέψη. Οι δύο θα έχουν ε, να κάνουν ε, με τον ρόλο των ενδιάμεσων δικηγόρων, τραπεζών κτλ. Και η άλλη έχει να κάνει με την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δανία, Γαλλία, κάτω και Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση αυτή, τους ερευνητέ μας, το προσωπικό των πολιτικών ομάδων που έμειναν εδώ μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ την Γραμματεία για τη στήριξή της επίσης και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος. Δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα, οπότε ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρίαση.